Ε, dear ε, Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, σας καλωσορίζω και θα ξεκινήσω καλησπερίζοντας όσους ήρθατε. Και μιας και υπάρχει διερμηνία θα μιλήσω τη μετρική μου γλώσσα, τα ελληνικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητέ φίλε και φίλοι, είναι με ιδιαίτερη χαρά που σα καλωσορίζω στο σημερινό μας, στη σημερινή μας συζήτηση, διάσκεψη. Είναι μια διάσκεψη μνήμης, τιμής και αγώνα αφιερωμένο στον ειρωνικό λαό της Παλαιστίνης και στη θλιβερή επέτειο των 50 χρόνων της κατοχής. Να σημειώσω ότι σε δύο μέρες, στις 29 Νοεμβρίου, είναι η διεθνή ημέρα αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό λαό. Μετά από μισό αιώνα κατοχής είναι προφανές ότι οι πολιτικές που έχουμε δεν συνεισφέρουν στην επίλυση του προβλήματος και την ειρήνη. Αυτό το έγκλημα συνεχίζεται εδώ και τόσα χρόνια με τη διεθνή κοινότητα να είναι απλώς παρατηρητής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε πως το Ισραήλ δεν λογοδοτεί για τα εγκλήματα του ενάντια στην ανθρωπότητα εδώ και 50 χρόνια παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και όλες τις διεθνείς συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Από το βήμα αυτό λαμβάνω ευκαιρία να επαναλάβω πως δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για να τεθεί ένα τέλος στην Ισραηλινή επιθετικότητα και να αποχρώσουμε επιτέλους του Ισραήλ να δεσμευτεί στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ. Επαναδετεπώνουμε πως αυτό το χρέος που απορρέει από τα καθήκοντά μας οφείλουμε να εργαζόμαστε αδιάλειπτα ώστε το Ισραήλ να σταματήσει να συμπεριφέρεται ως χώρα υπεράνω όλων των νόμων. Η επίλυση του Παλαιστινιακού και συνεπακόλουθα η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος και το κλειδί για να υπάρξει ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και να μπορέσουν όλοι οι λαοί της να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια. Δυστυχώς εδώ και 50 χρόνια οι πολιτικές του Ισραήλ παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα προκαλώντας τεράστια δεινά στους Παλαιστίνιους. Η βαρβαρότητα της Ισραηλής στρατιωτικής μηχανής συγκλονίζει κάθε φορά και περισσότερο. Σαν την προσωπία του Ευρωκοινοβουλίου με την Παλαιστίνη, είδαμε από κοντά στις επισκέψεις μας τις παράνομες πρακτικές του Ισραήλ. Κατεδαφίσεις οικισμό, σχολείο, σπιτιό, διοικητική κράτηση, δίκες και φυλακίσεις παιδιών και επιθέσεις στον άμαχο πληθυσμό. Παλαιστίνοι κρατούμενοι παραμένουν στι φυλακέ του Ισραήλ κατά παράβαση του άρθρου 49 τη 4 Διακρατική Συνθήκη τη Γενέβη, το οποίο απαγορεύει ρητά στην κατοχική δύναμη να μεταφέρει κρατούμενου μακριά από τι αιστείε του και τι οικογένειέ του. Το Συμβούλιο Ασφαλεία των Εθνών επίση έχει επανειλημμένα κηρύξει του Ισραηλινού υπηκισμού παράνομου. Χαρακτηριστικά είναι τα ψηφίσματα 465 και 2334 του Συμβουλίου Ασφαλεία, τα οποία διευκρινίζουν ότι ανοίγουν εισαγωγικά οι πολιτικοί και οι πρακτικέ επικισμοί του Ισραήλ στα κατεχόμενα αποτελούν ένα σοβαρό εμπόδιο στην επίτευξη μια συνολική, δίκαιη και μόνιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ενώ απευθύνουν κάλεσμα στο Ισραήλ να διαλύσει του υφιστάμενου οικισμού. Ακόμη, το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ήδη από τον Ιούλιο του 2004, έκρινε ότι ανοίγουν εισαγωγικά Ισραηλοί επικισμοί στα Παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένη και τη Ανατολική Ιερουσαλήμ, είναι παράνομοι. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Συνεπώ, η διεθνή κοινότητα ορίζει τερματισμό τη κατοχή και των παράνομων πρακτικών τη. Αντί αυτού, εδώ και 50 χρόνια το Ισραήλ επεκτείνει του παρόμοιου οικισμού στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτή η διαρκή επέκταση των επικισμών υπονομεύει κάθε ειρηνευτική προσπάθεια για την επίτευξη λύση δύο κρατών ταυτόχρονα παραβιάζει συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων που ζουν εκεί. Η δίμευση γη, η εκδίωξη, οι ανεξέλεκτε διακρίσει και οι ανέτε επιθέσει αποτελούν μέρο τη καθημερινότητα του λαού τη Παλαιστίνη. Ο στόχο είναι ένα. Ο κατακαιρματισμό του Παλαιστινιακού εδάφου, χωρίζοντα την ίδια ώρα γεωγραφικά του Παλαιστίνιου, που βρίσκονται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, σε δυτική όχθη, αλλά ε, και απομόνωση τη λωρίδα τη Γάζας. Οι κατάφερε παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Παλαιστινίων από τι Ιρανέ κατοχικέ δυνάμει συνεχίζονται. Η κατοχή εξευτελίζει και καταπιέζει καθημερινά την ανθρώπινη ύπαρξη στο καθεστώ του φόβου και τη καταπίεση. Το Ευρωκοινοβούλιο πολλέ φορέ σε ψηφίσματα του κατάγγειλε την επέκταση των επικισμών. Καταδίκασε τι κατεδεφάσει των Παλαιστινιακών υποδομών που πραγματοποιεί το Ισραήλ και ζήτησε την αναγνώριση ενό ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτου. Δεν μπορεί να υπάρξει μια λύση δύο κρατό χωρίς δύο κράτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη οφείλουν και πρέπει να αναγνωρίσουν την Παλαιστίνη ως κράτος. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε κάνει το μέρος που μας αναλογεί. Η διεθνή κοινότητα πρέπει να εφαρμόσει άμεσα το ψήφισμα 2334 τη Βουλή Ασφαλεία του ΟΗΕ, κάνοντα ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ των εδαφών του κράτου του Ισραήλ και των εδαφών που είναι κατεχόμενα από το 1967. Άρα Ολοκληρώνω να πω ότι ολοκληρώνοντα ζητούμε τη δημιουργία ανεξάρτητου κυρίαρχου και βιώσιου Παλαιστινιακού κράτου στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε να τερματιστεί ο απάνθρωπο αποκλεισμό τη Γάζα, να κρεμιστεί το παράνομο τείχο τη ντροπή που έστησε το Ισραήλ στη Δυτική να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι πολιτικοί, ε, Παλαιστίνοι πολιτικοί κρατούμενοι και να εξασφαλιστεί η επιστροφή των Παλαιστίνων προσφύγων όσο ορίζουν οι σχετικέ αποφάσει του ΟΗΕ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, είναι με μεγάλη χαρά που είδαμε την υπογραφή συμφωνία συμφωνίωση μεταξύ Χαμά και Φατάχ στον Κάιρο. Μια συμφωνία που ευελπιστούμε να τερματίσει τη μακρόχρονη ρήξη ανάμεσα στι δύο κύριε Παλαιστινιακέ οργανώσει. Θα παρακολουθούμε τι εξελίξει και αναμένουμε να οδηγήσει σε μια κυβέρνηση εθνική ενότητα, η οποία να έχει την ευθύνη και στη διδιώχθη και στη λωρίδα τη Γάζας και να δούμε να πραγματοποιούν όπως είναι και η συμφωνία εκλογές για όλα τα θεσμικά όργανα στην Παλαιστίνη, ενώ έχει οριστεί ότι μέχρι το τέλος του 2018 θα πραγματοποιηθούν αυτές οι εκλογές. Αγαπητοί φίλοι, σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε να στείλω από το βήμα αυτή τη διάσκεψη το μήνυμα αλληλεγγύη και προ τι φιλενικέ δυνάμει εντό του Ισραήλ. Ιδιαίτερα του Παλαιστίνου Άραβε πολίτε του Ισραήλ, οι οποίοι υφίστανται περιορισμών των πολιτικών του ελευθεριών καταπάτηση των δικαιωμάτων τους στη βάση πρακτικών apartheid που εφαρμόζει το Ισραήλ. Η αντιπροσωπεία των σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Παλαιστίνη στηρίζει έμπρακτα τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Καλούμε συστηματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάψει να τηρεί την μια αναπαράδεκτη πολιτική των ίσων αποστάσεων του Παλαιστινιακού. Το Ισραήλ παραβιάζει συστηματικά και βάνασα το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, με το Ισραήλ, το άρθρο 2 που αναφέρεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητούμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει δράση, να γίνει πρωταγωνιστικός ε, παράγοντας στην επίλυση του Παλαιστινιακού ζητήματος και να ασκήσει άμεσα πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τον επικισμό, να άρει την καρτοχή και να δημιουργηθεί σε έναν οδικό χάρτη για την ειρήνη και για τη λύση δύο κρατών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάσσονται στεναρά υπέρ μια λύση δύο κρατών ω το μόνο τρόπο για επίδεξη ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ε, σήμερα έχουμε αρκετού ε, ε προσκεκριμένου, επιφανεί, με ανάμειξη σε αυτόν τον ρόλο. Πριν όμω να μπούμε στη συζήτηση ε, των δύο ε, πάνελ που έχουμε, θα ήθελα να δώσω τον λόγο πρώτα στον πρέσβη της Παλαιστίνης για ένα πολύ σύντομο χαιρετισμό ε, τον έντιμο από απ τα Λαραχήμ Αλφάρα ε, να του δώσω λόγο για μια, ένα σύντομο χαιρετισμό. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Νεοκλή Σιλικιώτη πρόεδρε της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές και εκπρόσωποι των διαφορών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εξοχότητες και διαπιστευμένοι διπλωμάτες στις Βρυξέλλες. Κύριε Σάμουν, ε, δικαία απεσταλμένη του Προέδρου Αμπάς, και κύριε Πρέσβευτά της Παλαιστίνης στην Αίγυπτο, επιτρέψτε μου Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη της αντιπροσωπείας των σχέσεων με την Παλαιστίνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργανώσατε αυτή την τόσο σημαντική διάσκεψη για να ε, θυμηθούμε τα 50 χρόνια κατοχής του Ισραήλ, της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Γνωρίζετε τον, ε, τον ερτασμό την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου που θα γίνει για τον ε, Παλαιστινιακό λαό. Οι Παλαιστίνοι και όλη η χώρα ε, γιορτάζουν αυτήν την ημέρα, διότι όπως ξέρετε πριν από 70 ακριβώς χρόνια, 29 Νοεμβρίου 1947, η συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε το ψήφισμα 181 το ψήφισμα αυτό του διαμελισμού, όπως το λέμε. Το ψήφισμα αυτό ορίζει να δημιουργηθούν στην Παλαιστίνη δύο κράτη. Το Ισραηλινό κράτος, το οποίο ιδρύθηκε και συνεχίζει να υπάρχει, ενώ το κράτος της Παλαιστίνης περιμένει ακόμα να δημιουργηθεί. Όπως γνωρίζετε, το 1967, 5 Ιουνίου του 1967, το Ισραήλ ξεκίνησε την κατοχή στο 22% του εναπομείναντος ιστορικού εδάφους της Παλαιστίνης, την ε, Δυτική Όχθη δηλαδή, την ε, Δυτική Ιερουσαλήμ την Ελλάδα της Γάζας. Κατά συνέπεια, πάνω από 6 εκατομμύριο ε, Παλαιστίνοι ζουν σε εξορία και σε καταβλισμούς προσφύγων και 400 Παλαιστινιακά χωριά εξαφανίστηκαν από το χάρτη. Κυρίες και κύριοι, 80 χρόνια πέρασαν από... 24 χρόνια πέρασαν από την υπογραφή της Συμφωνίας του Όσλο, τα οποία μετά από 5 χρόνια προέβλεπαν τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης, όπως και τη διευθέτηση των ε, θεμάτων για το καθεστώς της Παλαιστίνης. Όμως έχουν περάσει 24 χρόνια και ακόμη περιμένουμε τη δημιουργία του κράτους μας. Από την άλλη, εμείς, οι Παλαιστίνοι, έχουμε αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ στα σύνορα του 1967 ενώ το Ισραήλ αρνείται ακόμη να αναγνωρίσει τα ίδια τα σύνορά του ε, και συνεχίζει να δημιουργεί επικισμούς ε, ε, με σε κατάφορη παραβίαση των διεθνών συμφωνιών και ψηφισμάτων καθώς και του διεθνούς δικαίου. Κυρίες και κύριοι, είναι στιγμή, είναι καιρός να δώσουμε τέρμα στην Ισραηλινή κατοχή. Η κατοχή αυτή είναι όνειδος για το Ισραήλ και για τη διεθνή κοινότητα. Η κατοχή αυτή αποτελεί μια κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του ε, κράτους δικαίου για το λαό μας. Κυρίε και κύριοι, η ειρήνη δεν χτίζεται από τη μία μόνο πλευρά. Παρόλα όσα έχουν γίνει, οι δυνάμεις κατοχής του Ισραήλ ε, συνεχίζουν να μην σέβονται τις δεσμεύσεις τους για τη λύση δύο κρατών και συνεχίζουν να επιβάλλουν την πολιτική του τετελεσμένου στο έδαφος της Παλαιστίνης και όλος ιδιαίτερο στην ε, κατοχή της Δυτικής Ιερουσαλήμ, της Ανατολικής Τη δυτική Ιερουσαλήμ. Το Ισραήλ απορρίπτει τι λύσει που προτείνονται ω τώρα με διπλωματικέ οδού και τι πρωτοβουλίε για την ειρήνη. Και επαναλαμβάνω, η ειρήνη δεν χτίζεται από τη μία και μόνο πλευρά. Δεν μπορούν μόνοι του οι Παλαιστίνοι να φτιάξουν την ειρήνη από τη στιγμή που πρέπει να υπάρχουν δύο πλευρές που συμφωνούν για να υπάρξουν συνθήκες ειρήνης. Το Ισραήλ με αυτή την κυβέρνηση, το Ισραήλ με αυτή την του Νετανιάχου δεν θέλει ειρήνη, είναι σαφές. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω απλώς αυτό που είπε ο πρόεδρός μας στο ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο κ. Σαμπάς. Και θα αναφέρω τα λόγια του. Ο κίνδυνος, ο κίνδυνος που πλησιάζει κατά του λαού μας και της ύπαρξής μας στο διεθνές προσκήνιο και την οικονομία καθώς και την πολιτική ε, στο έδαφος μας που απειλεί την ασφάλεια και την ειρήνη στο ε, στη δική μας περιοχή και στον κόσμο, μας αναγκάζει να αναλάβουμε μέτρα που θα ε, υποχρεώσουν την δύναμη κατοχής να ε, πάυσει την κατοχή της. Πρέπει να εξεύρουμε ανελακτικές λύσεις που θα διαφυλάξουν τα δικαιώματά μας και θα προστατεύσουν την γη μας και τον λαό μας από τις πρακτικές apartheid που εφαρμόζει το Ισραήλ η δύναμη κατοχής. Τέλος του παραθέματος. Κυρίες και κύριοι, εάν μιλήσω για τα εσωτερικά προγράμματα των Παλαιστινίων, θα πρέπει να αναφέρω το εξής. Το πρόγραμμα για την οικοδόμηση της χώρας μας προχωράει σταδιακά για την οικοδόμηση εθνικών θεσμών. Έχουμε θεσπίσει υποδομές, βασικές υποδομές για τη χώρα μας, πράγμα που γίνεται σε συμφωνία με την αρχή του κράτους δικαίου που θέλουμε να εδραιώσουμε ε, καθώς επίσης και το ρόλο των γυναικών και των νέων. Ταυτόχρονα επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την εθνική συμφιλίωση ώστε να δοθεί τέρμα στους διαχωρισμούς και τις διενέξεις και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια κυβέρνηση εθνικής συμφιλίωσης και υπό την Αγία τη Αιγύπτου και να ε, βρούμε λύσει και για την Λωρίδα τη Γάζας και για την Δυτική Όχθη ώστε να εδρεωθεί μία μόνη αρχή, μία μόνη κυβέρνηση και, νόμιμα, ε, ε, και νόμιμες οδοί επίλυσης των διαφορών. Κυρίες και κύριοι, χαιρετίζουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της και παροτρύνουμε όλου να συνεχίσουν άοκνα τι προσπάθειέ του για να δοθεί τέρμα στην Ισραηλινή κατοχή. Στο κράτο τη Παλαιστίνη να δοθούν σάρκα και οστά και επιτέλου να γίνει πραγματικότητα η λύση των δύο κρατών. Για να γίνει σεβαστή η αρχή τη ισότητα και τη δικαιοσύνη, καλούμε τις χώρες που ακόμη δεν έχουν αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης να το πράξουν και μάλιστα αμέσω. Νομίζω ότι τώρα ή ποτέ έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θέλω επίση να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλου του Ευρωπαίου πολίτε για την στήριξή του, τη διαρκή του υποστήριξη προ τον Παλαιστινιακό λαό σε αυτά τα χρόνια δημιουργίας του κράτους, εδραίωσης ε, και οικοδόμησης της οικονομίας μας. Ο λαός μας σας είναι ευγνώμων. Για να ολοκληρώσω, να ευχαριστήσω, αγαπητοί φίλοι, από τα βάθη της καρδιάς μου όλους σας για την ελληνική που επιδεικνύεται προς τον Παλαιστινιακό λαό για το δίκαιο ε, ε, αγώνα μας και για την ε, δέσμευσή σας να μείνετε στο στατόπεδο της δικαιοσύνης και της ειρήνης. Ελπίζω ότι σύντομα θα έρθει η μέρα που θα δοθεί τέρμα στην Ισραηλινή κατοχή και όπου ο λαός μας θα είναι πια ανεξάρτητος και ελεύθερος στη χώρα του. Με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και εκεί να μπορέσουμε και να σας υποδεχθούμε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Thank ε, Σας ευχαριστώ κύριε Αλφάρα, σας ευχαριστώ πρέσβη και τώρα Θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους από την Παλαιστίνη. Ε, θα, θα δώσω το λόγο στον ειδικό απεσταλμένο του Προέδρου Αμπάς, τον κύριο Γιούνεσάμ. مع فلسطين في البرلمان الأوروبي السادة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 κύριοι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, κύριοι και κυρίες διπλωμάτες, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, κύριε Αμπραχήμ Ιφτά. يسرني أن ألتقي بكم هنا في بروكسل لأنقل لكم تحيات فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وأركان القيادة الفلسطينية وتحيات شعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي الشتات والمهاجر الذي يتطلع إلى عونكم ومساعدتكم له في تحقيق استقلاله وحريته It's a pleasure to... Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι ενώπιόν σα σε αυτή τη συνεδρίαση της, των Βρυξελών και σας διαμηνύω τα χαιρετίσματα του κυρίου Μαχμούτα Αμπάς, πρόεδρου της Παλαιστίνης, και τους χαιρετισμού του Παλαιστινιακού λαού που βρίσκεται υπό κατοχή, ο οποίος περιμένει τη βοήθεια και τη στήριξή σας για να εξασφαλίσει την ελευθερία και την ανεξαρτησία του. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της ε, Επιτροπής για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη, που οργάνωσαν αυτή την ε, ε, συνεδρίαση για τα 50 χρόνια κατοχής. يصادف بعد يومين من هذا اليوم وهو يوم التاسع والعشرين من نوفمبر سأورد لكم أجزاء من رسالة فخامة رئيس دولة فلسطين بهذه المناسبة. Όπως ξέρετε κυρίες και κύριοι, στις 28 Νοεμβρίου, σε δύο μέρες, έχουμε τη Διεθνή ημέρα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. Επ' λοιπόν, θα ήθελα να σας μιλήσω ε, για ένα κομμάτι της επιστολής του κυρίου Μαχμού Ταμπάς. اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 والمعروف بقرار التقسيم والذي نص على أن تنشأ في فلسطين دولتان πριν από 70 χρόνια, τον Νοέμβριο, η Γενική Συνέλευση του, ΟΗΟ, ΟΗΕ εξέδωσε το ψήφισμα 181, το ψήφισμα για τη διαίρεση, όπως είναι γνωστό, που είπε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν δύο κράτη στην ιστορική Παλαιστίνη. Ε, بل إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في بلادنا قامت عام 1948 بعملية اقتلاع لنصف الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده من دياره بقوة النار والإرهاب One state. Το ένα κράτος δημιουργήθηκε με βάση αυτό το ψήφισμα. Το 1948 δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ και ρίζωσε εκείνο, ενώ ξερίζωσε τους Παλαιστίνιους παράλληλα που ζούσαν εκεί. Έτσι ξεκίνησε η Παλαιστινιακή ε, Διασπορά. Σήμερα ελέγχουν πάνω από το έδαφο που θα έπρεπε να ελέγχουμε βάση το ψήφισμα αυτό της διαίρεσης. والبالغة 22% من أرض فلسطين التاريخية. Το 1967 το Ισραήλ κατήχε το κατέλαβε το υπόλοιπο 22% της ιστορικής Παλαιστίνης, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας. Which is the West Bank and Gaza Strip and East Jerusalem. وترتب على ذلك أن أكثر من 6 مليون فلسطيني يعيشون في ديار اللجوء والشتات Έξι εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη διασπορά εξαιτία αυτή τη κατάσταση. Και αυτό οδήγησε στην καταστροφή 418 πόλεων και χωριών στην Παλαιστίνη. Πριν από 70 χρόνια, αμφισβητήθηκε η ύπαρξη των Παλαιστίνιων στη γη τους. Και εδώ και 50 χρόνια υπάρχει κατοχή και στα υπόλοιπα Παλαιστινιακά εδάφη. Οι Παλαιστίνοι ακόμη περιμένουν τη δικαιοσύνη να αποκατασταθεί από τη διεθνή κοινότητα. Βλέπουμε πάντα με θετικό μάτι όλες τις πρωτοβουλίες που προωθούνται για την ειρήνη. Ακόμα περιμένουμε να γίνουν περισσότερα πράγματα για να πετύχουμε το σκοπό μας. مع المبادرات والجهود التي بذلت ولا زالت تبذل وقد ضحى شعبنا بعشرات آلاف الشهداء والجرحى ويتعرض مئات الآلاف من أبنائه في وطنهم فلسطين لأشكال العذاب العذابات والقمع والتنكيل والاعتقال في سجون دولة إسرائيل القائمة بالاحتلال لأرض دولة فلسطين. And all, through all this time, as you all... Όλα αυτά τα χρόνια, όπως ξέρετε, οι Παλαιστίνοι θυσιάστηκαν κατά δεκάδες, εκατοντάδες, κατά χιλιάδες και χιλιάδες Παλαιστίνοι υφίστανται τα δεινά και τις ταπεινώσεις της κατοχής από το κράτος του Ισραήλ που κυριαρχεί τα Παλαιστινιακά, στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και απαγορεύει και δεν δίνει στους Παλαιστίνιους τα πιο θεμελιώδη, τα πιο βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουν το δικαίωμα να... στην αυτοδιάθεση. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν αυτό το δικαίωμα. και να απολαμβάνουν την ανεξαρτησία τους στα εδάφη τους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Κυρίε και κύριοι, 24 χρόνια πέρασαν από την υπογραφή των συμφωνιών του Όσλου. που υποτίθεται θα οδηγούσε σε έναν εξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος πέντε χρόνια μετά την υπογραφή. και θα επέλυε και διάφορα άλλα θέματα που παρέμεναν εκκρεμή και που, είχαν, και που αναφερόταν στις συμφωνίες. Από πλευράς μας αναγνωρίσαμε την παρουσία του Ισραήλ και τα σύνορα του 1967. Το Ισραήλ αρνείται να αναγνωρίσει τα σύνορα αυτά ως τελικά σύνορα του Ισραήλ και συνεχίζει την κατασκευή των επικισμών στα κατεχόμενα εδάφη μας. Με αυτόν τον τρόπο αρνείται την ανεξαρτησία του κράτους μας παραβιάζοντας κατάφορα το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή ψηφίσματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρνούμενο τη λύση των δύο κρατών και κάνει ό,τι μπορεί για να απαγορεύσει την υλοποίηση αυτών των λύσεων. لقد حان الوقت لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين والذي يشكل وصمة عار في بل إنه عدوان غاشم على الحرية وحرية شعبنا وحقوقه ولا يمكن للمجتمع الدولي مواصلة سياسة كيل بمكيالين والتعاطي بمعايير مزدوجة Κυρίε και κύριοι, είναι και καινή ώρα να τεθεί τέλο στην Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Αυτή η κατοχή αποτελεί ντροπή για το Ισραήλ και τη διεθνή κοινότητα και για οποιονδήποτε υποστηρίζει την λύση αυτή, την κατάσταση αυτή. Η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτά τα διπλά μέτρα και σταθμά. στηρίζοντας την Ισραηλινή κατοχή. وتمكين شعبنا من تقرير مصيره على أرضه ونيل حريته والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمته القدس الشرقية على حدود 67 The political and η πολιτική τα πολιτικά προβλήματα, η, τα ανθρώπινα βάσανα για την κατοχή είναι ευθύνη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κουαρτέτου του ΟΗΕ και του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτοί θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτω ώστε οι Παλαιστίνοι να έχουν το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, να έχουν ανεξάρτητο κράτος στα εδάφη που κατέχουν από το 1967 οι Ισραηλοί και θα πρέπει να του δοθεί το δικαίωμα να έχουν πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. وسينزع من التنظيمات الإرهابية الذرائع والمبررات التي تستخدمها لبث أفكارها الظلامية The end of the Israeli... Το τέλος της Ισραηλινής ε, κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη θα βοηθήσει στο να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Αυτές οι οργανώσεις εξαπλώνουν τις σκοτεινές ιδέες τους και βρίσκουν και θεωρητική υποστήριξη στις δολοφονίες αθώων ανθρώπων. Είμαστε μαζί με την διεθνή κοινότητα. Θέλουμε να αντιμετωπιστεί η διεθνής τρομοκρατία και να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Κυρίες και κύριοι, ο πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς, ο πρόεδρος της Παλαιστίνης, επιβεβαίωσε κατ' επανάληψη ότι ο βασικός μας στόχος είναι η ειρήνη. η Παλαιστίνη έκανε ό,τι μπορούσε για να υλοποιηθεί ε, η ειρήνη. Και έχουμε υποστηρίξει την Αραβική Πρωτοβουλία για την Ειρήνη. Υλοποιήσαμε επίσης όλες τις προϋποθέσεις του Αμερικανικού Οδικού Χάρτη με βάση την, την Ειρηνευτική Πρωτοβουλία. Υποστηρίξαμε και όλες τι υπόλοιπε πρωτοβουλίε που προωθούν ε, την ειρηνευτική διαδικασία και τη λύση των δύο κρατών. Εδώ συμπεριλαμβάνεται η γαλλική πρωτοβουλία, η πρωτοβουλία του Πρόεδρου Πούτιν, του Κινέζου Προέδρου και οι προσπάθειες του Ντόναλτ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία που θα θέσει τέλος ε, στη σύγκρουση με βάση τις διεθνείς, τα διεθνή ψηφίσματα και τη λύση των δύο κρατών. Παρά, το, παρά τις προσπάθειες αυτές, το Ισραήλ επιμένει συνεχίζει την κατοχή και δεν συμμορφώνεται με τη λύση των δύο κρατών. Παρά τις προσπάθειες αυτές, το Ισραήλ συνεχίζει το status quo στα Παλαιστινιακά εδάφη, στην κατεχόμενη Ισραηλ, Ιερουσαλήμ και συνεχίζει να οικοδομεί επικο, επικισμούς αρνούμενο την, α, τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες. Η ειρήνη δεν μπορεί να οικοδομηθεί από τη μία πλευρά μόνο. And all the οι πρακτικές του Ισραήλ εντός των Παλαιστινιακών εδαφών είναι κενές και δεν έχουν καμία ε, νομική ή ηθική βάση. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αυτές τις πρακτικές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Στα ιερά εδάφη για το Ισλάμ και για το χριστιανισμό και να διατηρήσει την ιστορική νόμιμη κατάσταση και καθεστώς ε, σε αυτά τα ιερά εδάφη, κυρίως ε, στο Ιερό Τζαμί. Επιβεβαιώνω αυτό που είπε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος Αμπάς στον ΟΗΕ. Ο άμεσος κίνδυνος που στοχεύει την παρουσία μας, τα δικαιώματά μας, τη διεθνή και πολιτική παρουσία μας στην ε, γη μας, απειλεί την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας και στον κόσμο. Πρέπει το Ισραήλ να, επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες του για τα αποτελέσματα της κατοχής. Και θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις για να διατηρηθούν τα εδάφη μας και τα δικαιώματα του λαού μας. Να αντιμετωπιστεί το apartheid που ασκεί το Ισραήλ στα εδάφη μας με τη βία και μέσω της κατοχής των εδαφών μας. Κύριε Πρόεδρε, ο, ο Πρόεδρος μάλλον προσέθεσε επίσης οι επιλογές μας για να συμμορφωθούμε με το διεθνές δίκαιο είναι ότι το διεθνές δίκαιο είναι η αναφορά μέσα στην... και μέσα στο, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου θα βρεθεί λύση, ε, μία λύση δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967. Υπάρχει υποστήριξη από εμά από προηγούμενες πρωτοβουλίες. Και λαμβάνουμε υπόψη μα τι προσπάθειες που καταβάλει ο πρόεδρος Τραμπ τα μέλη του κουαρτέτου και η διεθνής κοινότητα, ούτω ώστε να υπάρξει μια ευκαιρία για να υπάρξει ιστορική συμφιλίωση και μια συμφωνία για τη λύση των δύο κρατών. Αν αυτές οι προσπάθειες αποτύχουν, τότε θα ασκήσουμε τα δικαιώματά μας είναι τα ίδια δικαιώματα που έχουμε με τους Παλαιστίνιους. Ανεξάρτητα από τη φυλή μας, από την προέλευσή μας, από το χρώμα μας, έχουμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα σε αυτά τα εδάφη. Εμείς, οι Παλαιστίνοι, οι μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τον Εβραϊσμό ως θρησκεία. Η βασική μας αντιπαράθεση είναι απέναντι στο Ισραήλ και στην απεικιοκρατική στάση του και στην οικοδόμηση των επικισμών που κυριαρχούν στο λαό μας και στα εδάφη μας ε, επί δεκαετίες. κυρίες και κύριοι, η κατάσταση εσωτερικά της Παλαιστίνης είναι μια κατάσταση που εξελίσσεται, οικοδομούμε τις απαραίτητες υποδομές στο Παλαιστινιακό κράτος, με βάση το κράτος δικαίου, μέσα στα πλαίσια μιας προσπάθειας ενίσχυσης των νέων και των γυναικών, Από την άλλη, προσπαθούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Την υποστήριξη της Αιγύπτου κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να υπερκεράσουμε τα εμπόδια που δημιουργούν προσκόμματα στην εθνική ενότητα και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στη Γάζα. Θέλουμε να υπάρξει μία αρχή στα Παλαιστινιακά εδάφη ε, με ένα δίκαιο. Επομένως, συνεχίζουμε τις επραγματεύσεις μας και με την κυβέρνηση της Γάζας και με την κυβέρνηση της Δυτικής Όχθης. حثها Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και ελπίζουμε ότι θα συνεχίζουν να υποστηρίζουν τις παλαιστινιακές προσπάθειες για να τεθεί τέρμα στην Ισραηλινή κατοχή να σταματήσουν οι επικισμοί και η απεικιοκρατική πολιτική του Ισραήλ και να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναγνωρίζουν το Ισραήλ να το αναγνωρίσουμε βάσει τα σύνορα του 1967 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και ζητούμε από όλα τα κράτη-μέλη να σταματήσουν οποιαδήποτε άμεση ή έμεση επαφή με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Γιατί είναι παράνομη.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 And θα ήθελα να ευχαριστήσω τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κάθε Ευρωπαίο για τη στάση του και την υποστήριξή του απέναντι στους Παλαιστινίους στην προσπάθειά του να οικοδομηθούν οι απαραίτητοι θεσμοί και η οικονομία του. Ελπίζουμε να ξέρετε ότι οι Παλαιστίνοι σέβονται την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους. من صميم قلبي على تضامنكم مع شعبنا وقضيته العادلة مثمنا عاليا جهودكم النبيلة والمخلصة لكل فرد منكم Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου από βάθους καρδίας για την αλληλεγγύη και στήριξή τους απέναντι στο παλαιριστινιακό λαό. Σας σέβομαι για τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλατε και που σας έδωσαν και το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη. Ελπίζω κάποια μέρα θα γιορτάσουμε το τέλος της Ισραηλινής κατοχής. Και ο λαός μας θα ζήσει ελεύθερος, ανεξάρτητος στη δική του χώρα με πρωτεύουσα την ε, Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ευχόμαστε μάλιστα αυτό να υλοποιηθεί πολύ σύντομα. ούτω ώστε να έχουμε και την τιμή να σας υποδεχτούμε στη χώρα μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γιουνεσάμ. Ειδική απεσταλμένη του Πρόεδρου Αμπάς. εκ μέρου όλη τη αντιπροσωπεία θέλω να εκφράσετε την αλληλεγγύη μα προ τον πρόεδρο Αμπά και τον ολόκληρο τον Παλαιστινιακό λαό. Ε, ανέκαθεν πιέζαμε για μια λύση ειρήνης, για μια δίκαιη λύση και τώρα θα καλέσω τον συνάδελφο Ιβο Βάικλ ε, που είναι μέλος της ε, αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη και πρώην υπουργό της Σλοβενίας να, λάβει το, να έρθει να προεδρεύσει. Με, θα ακούσουμε τον κύριο Χάμεμπεργκ, τον κύριο Λίνκ και την κυρία Αζάροβα στο πάνελ. Ladies and gentlemen, it is, it is an honor for me to... Κυρίες και κύριοι, είναι τιμή μου να προεδρεύω σε τέτοιο πάνελ με τέτοιους επίτιμους, ε, ξέχοντες μάλλον προσκεκλημένους και παρεμβαίνοντες. Θέλω να σας καλωσορίσω όλους, ειδικά όσους ήρθατε από την Παλαιστίνη και να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μας τον κύριο Σιλικιώτη ο οποίος είναι ο ίδιος ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. και παρακολουθεί το θέμα του ανεξάρτητου κράτους και του κυρίαρχου κράτους της Παλαιστίνης ε, με ιδιαίτερη ε, ενεργητικότητα σε αυτό το κοινοβούλιο. Ε, ό,τι συζητούμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο έχει σκοπό να συνεισφέρει στην ε, κατανόηση από την πλευρά του λαού της ε, Παλαιστίνης και τη συνεννόησή του με το λαό του Ισραήλ. Δεν είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ. Είμαστε υπέρ της ειρήνης στην περιοχή. Και προκειμένου να βρεθεί μια λύση που να καλύπτει και τις δύο πλευρές και τα δύο έθνη που συγκατοικούν στην Παλαιστίνη. 50 χρόνια κατοχής υπόθηκε ήδη, είναι η επέτειος που γιορτάζουμε αλλά ακόμη και ένας μήνας κατοχής θα ήταν ε, βάρος και ο οδυνηρό για όσους αναγκάζονται να υποστούν την κατοχή. Νομίζω το μήνυμα αυτής της διάσκεψης θα πρέπει να είναι ας δώσουμε στην ειρήνη μια ευκαιρία στη Μέση Ανατολή. Διότι αν δεν υπάρξει δίκαιη λύση εάν δεν υπάρξει ειρηνική λύση, θα οδηγηθούμε στην καταστροφή. Πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου να το επαναλαμβάνω αυτό διαρκώς, αλλά ως φίλος της ειρήνης και φίλος όσων κατοικούν στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, είχα την τιμή να τους συναντήσω και τους μεν και τους δε επανειλημμένους. Και γνωρίζω ότι οι άνθρωποι και των δύο εθνών την ειρήνη θέλουν. Θέλουν να ζήσουν ειρηνικά. Δυστυχώς όμως η πολιτική και τα πολιτικά πράγματα οδηγούν την διαδικασία σε άλλη κατεύθυνση. Αυτό λοιπόν το οποίο θα προσπαθήσουμε να συζητήσουμε σήμερα, αυτό ακριβώς το γεγονός έχει σκοπό να υπογραμμίσει. Παρόλα αυτά, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο ως θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναλάβουν έναν ενεργό ρόλο στη δικασία της Ειρήνη. και να ε, γίνει αυτός ο σκοπός μας με περισσότερα κίνητρα και προσπάθειες. Δεν γίνεται απλώς να επαναλαμβάνουμε στα λόγια τις ίδιες τοποθετήσεις, τα ίδια επικριτικά σχόλια την ίδια θλίψη που, και δυσαρέσκεια για όσα συμβαίνουν στην Παλαιστίνη. Με συγχωρείτε που έκανα κατοχή στο μικρόφωνο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Είμαι συντονιστής αυτού του πάνελ, αυτών των επιτήμων εξεχόντων προσκεκλημένων και κατά πρώτο να δώσω το λόγο στον κύριο Μάικλ Λίνκ ο οποίος είναι ειδικό απεσταλμένο στο ΙΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα κατεχόμενα της Παλαιστίνη και είναι ε, καθηγητής στο, στη νομική στο Western University του Λονδίνου ε, στο Οντάριο του Καναδά. Ε, θα επαναλάβω, ε, καθώς παρουσιάζω για τους προσκεκλημένους μας, ότι αναλυτές και μελετητές προσκεκλημένοι είναι εδώ όσοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά εδώ και χρόνια και είναι αφοσιωμένοι φίλοι της διαδικασίας ειρήνης στην περιοχή. Κύριε Λίνκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση και τη σύσταση. Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μπορώ να απευθυνθώ στο Ευρωκοινοβούλιο για ένα θέμα τόσο σημαντικό γνωρίζετε το θέμα του Ισραήλ και της Παλαιστίνης απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση σε, πολλά, σε πολλούς τομείς της εξωτερικής της πολιτικής και ελπίζω οι σημερινές συζητήσεις να βοηθήσουν να εμβαθύνετε και να προχωρήσετε το πολύ καλό έργο που ήδη κάνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα την τιμή τον Οκτώβριο να δημοσιεύσω την τρίτη μου έκθεση στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την παρουσίασα και επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο θέμα το νομικό πλαίσιο της κατοχής. Η ουσία της δουλειά μου, της έκθεσης αυτής, είναι ότι χρειαζόμαστε μια νέα προσέγγιση, ένα νέο νομικό πλαίσιο, έναν νέο τρόπο για να μπορέσουμε να μελετήσουμε πού οδεύει αυτή η κατοχή. Η έκθεση που έχω συντάξει αιτιολογείται από το γεγονός ότι υπάρχει μια ε, ένα διέξοδο στην κατοχή και ότι οι, οι Παλαιστίνοι διεκδικούν την ειρήνη, το ίδιο και οι Ισραηλινοί. Είναι πολλές οι ιδέες που ακούγονται και έχουν δοκιμαστεί, αλλά οι περισσότερες έχουν ήδη αρχίσει να χάνουν την ενέργειά τους. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν την, ουσία, των βασικών σημείων της εκθεσής μου το προηγούμενο μήνα. Όπως πολλοί από εσά τα γνωρίζετε και το υπενήχθησαν και οι ομιλητές του εισαγωγικού πάνελ, τον Ιούνιο του 1967 το Ισραήλ άρχισε να κατέχει ή τέλος πάντων να περνάει σε επικισμό της Δυτικής Ιερουσαλήμ και της Λεωρίδας της Γάζας. Γιορτάζουμε τα 50 χρόνια και σύμφωνα με τα στοιχεία του Ερυθρού Σταυρού αυτή είναι η μακρύτερη σε διάρκεια στρατιωτική κατοχή στον κόσμο. Ε, η διεθνής κοινότητα ε, θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι η δύναμη κατοχής. Αυτό επιβεβαιώθηκε από το ψήφισμα του Συμβουλίου Ειρήνης 2334 ε, τον περασμένο Δεκέμβριο και από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με το ψήφισμα 7196 και αυτό το περασμένο Δεκεμβρίου το εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της κατοχής. Τα βασικά όργανα αυτά είναι ο κανονισμός της Χάγης, το πρωτόκολλο του 1967 και ούτω καθεξής και εδώ συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις για τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και το διεθνέ ποινικό δίκαιο. Όλα αυτά θα πρέπει να διέπουν την διαδικασία κατοχής. Το Ισραήλ μόνο αυτό από τα μέλη του ΟΗΕ αρνείται να αναγνωρίσει την κατάσταση αυτή ως κατάσταση κατοχή. Και αρνείται να αναλάβει τι ευθύνε του ω ε, δύναμη κατοχή. Κατά τη... κατά... Καθώς εξ όσων μάλλον γνωρίζω, είναι το μόνο κράτο που δεν αναγνωρίζει το καθεστώ του κράτο κατοχή. Τα τελευταία 50 χρόνια η διεθνής κοινότητα θεωρεί το Ισραήλ ως νόμιμο ε, κάτοχο των κατεχομένων ε, της Παλαιστίνης. Υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου όμως εδώ, όπως οι επικισμοί, η οικοδόμηση τείχους, παλαιστινιακά εδάφη, η προσάρτηση της ε, Ανατολικής Ιερουσαλήμ το 1967-1980 και μια σειρά από παραβιάσεις ανθρωπινών δικαιωμάτων. Το ερώτημα που θέτω στην έκθεσή μου, ερώτημα που θέλω να θέσω και σε εσά σήμερα, είναι. Μπορεί ένας ένομος κάτοχος να ξεπεράσει κάποιες απαγορευτικές γραμμές, μια, ένα όριο και να γίνει παράνομος ε, κατέχων. Εάν ισχύει αυτό, ποιες θα είναι οι συνέπειες. Δεν ε, αλλάζει κάτι με το ότι μιλάμε για μια κατοχή 50 ετών. Ένας ένομος κατέχων που ξεπερνάει τα όρια και γίνεται παράνομος, ανα πάσα στιγμή, είτε είναι στην αρχή της κατοχής είτε προς το τέλος, είτε πριν από 20-30 χρόνια, δεν αλλάζει κάτι. Και ω ειδικό απεσταλμένο στην έκθεση αυτή τονίζω ότι δεν έχει σημασία πότε ακριβώ συνέβη αυτό. Σημασία έχει ότι εδώ και 50 χρόνια πρέπει να εξετάσουμε αν ξεπεράστηκε αυτό το όριο από το Ισραήλ. Το Διεθνέ Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και αν δείτε τα βασικά έγγραφα και εργαλεία που το ε, αναλύουν, δεν δίνει συγκεκριμένη απάντηση σε αυτό. Όμως μπορούμε να βρούμε απάντηση αν εξετάσουμε τα γενεσιουργά έτα και τα θεμέλια του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό σας προτείνω να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εξίβρα τέσσερα, τέσσερις σημαντικές αρχές επί των οποίων μπορούμε να βασιστούμε, που μπορούμε να ε, εξάγουμε, εξεγάγουμε από το ε, Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Δεν αφορά ειδικά το Ισραήλ, αλλά οποιαδήποτε ένοπλη μακράς διάρκειας κατοχή. Για να δούμε κατά πόσο ένα ένομος κατέχων γίνεται παράνομος. Δεν χρησιμοποιώ τον όρο παράνομη κατοχή. Η κατοχή υπό το Διεθνέ Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θεωρώ ότι είναι ουδέτερο όρο. Το ερώτημα είναι αν ο κατέχον, αυτό που χειρίζεται, που πραγματοποιεί την κατοχή, από ένομος κατέχον έχει περάσει στο καθεστώ της παρανομία. Το πρώτο λοιπόν από τα τέσσερα σημεία που θέλω να σας επισημάνω είναι ότι είναι πολύ σαφής ο ορισμός στο Διεθνέ δίκαιο. Ότι ο κατέχον δεν έχει κανένα δικαίωμα σε κανένα από τα κατεχόμενα εδάφη. Από το 1945 έχουμε ξεπεράσει την αρχή της κατάκτησης. και βλέπουμε ότι στο ψήφισμα του 2334, θα το δείτε στην αρχή του PowerPoint μου, ότι είναι απαράδεκτη η ε, προσάρτηση εδαφών με τη βία. Αυτή είναι τουλάχιστον η 8η φορά που το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εγκρίνει ένα τέτοιο ψήφισμα με τέτοια φρασιολογία σε ψήφισμά του σε σχέση με την Ισραηλινή κατοχή Παλαιστινιακών ή άλλων αραβικών εδαφών. Αυτό είναι και μέρος του εθιμικού διεθνούς δικαίου, όπως ε, οι αρχές του διεθνούς δικαίου που εγκρίθηκαν ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ ομόφωνα το 1970 δεν μπορεί να υπάρχει προσάρτηση εδαφών με τη βία και να θεωρείται νόμιμη. Η προσάρτηση εδαφών έγινε σε πόλεμο αμυντικό, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ για τον πόλεμο το 1967, ή σε πόλεμο επίθεσης. Εγώ ε, θα εισηγηθώ ότι δεν χρειάζεται να απαντηθεί αυτό το ερώτημα για να δούμε τι έγινε το 1967, ε, ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι η επιχειρηματολογία του Ισραήλ είναι σωστή και ότι προσάρτησε τα Παλαιστινιακά εδάφη το 1967 επειδή είχε ένομο πόλεμο άμυνας κατά των Παλαιστινίων αυτοάμυνα, η οποία όμως παρόλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν ξεπέρασαν το απαγορευτικό όριο και δεν παραβίασαν αρχές του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν πρώτη αρχή ήταν η αρχή της μη προσάρτησης. Δεύτερη αρχή. Η κατοχή είναι, νομι... είναι διαρκής ή προσωρινή. Ο κατέχον ε, απαιτείται να επιστρέψει τα εδάφη στον λαό του οποίου... στον οποίο ανήκαν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Με άλλα λόγια, ε, η κατοχή μπορεί να είναι προσωρινή. Δεν μπορεί να είναι παορίστο, ούτε να είναι μόνιμη. Αυτό το ε, βλέπουμε σε απολυταρχικά σχόλια, σε σχόλια ε, ε, που έγιναν τα τελευταία χρόνια η αμερικανική κατοχή της Ιαπωνίας μετά το 1945 λόγω χάρη, η, κατοχή της Δυτικής Γερμανίας από τους συμμάχους μετά το 1945, η, Αμερικανική, ο η αμερικανική, μάλλον υπό η αμερικανική αιγίδα ε, κατοχή του Ιράκ από τις συμμαχικές δυνάμεις πρόσφατα. Αυτές οι αρχές που διέπουν την κατοχή οδήγησαν σε μια διάρκεια το πολύ δεκαετίας. Το πολύ δεκαετίας εδώ μιλάμε για μια κατοχή που συνεχίζεται για 50 και να σας θυμίσω ότι το 1980, τον Ιούνιο του 1980, επ' ευκαιρία της 30ης επαιτίου από την αρχή της κατοχής, ε, η συνέλευση του ΙΕΝ έκρινε ψήφισμα που ήδη τότε εξέφραζε το κατά πόσο είναι ήδη ανησυχητική μεγάλη διάρκεια της κατοχής του Ισραήλ. Ήταν το ψήφισμα 47-86. Ε, Αυτό το ψήφισμα του 80 ε, επαναλαμβάνει, και θα παραθέσω εδώ το κείμενο του ψηφίσματος, ότι η ε, επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η μακροσχελέστατη αυτή κατοχή των αραβικών ανταφών από το Ισραήλ είναι αντικείμενο δυσαρέσκειας και θα πρέπει το Ισραήλ να συμμορφωθεί με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. 37 χρόνια πριν, περίπου ένα τέταρτο της διάρκειας της κατοχής. Ήδη τότε το Συμβούλιο Ασφαλείας και Γενική Συνέλευση εξέφραζαν ανησυχία για τη μεγάλη διάρκεια της κατοχής και την άρνηση, την ε, συστηματική άρνηση του Ισραήλ να ακολουθήσει και να συμμορφωθεί με τι επιταγέ των ψηφισμάτων τη Γενική Συνέλευση και του Συμβουλίου Ασφαλεία. Τρίτη αρχή σε σχέση με την κατοχή και το κατά πόσο είναι ένομη ή παράνομη είναι το εξής. Ότι ο κατέχων κατά τη διάρκεια όλη τη διάρκεια τη κατοχής πρέπει να δικεί ε, κατά το συμφέρον του κατεχόμενου λαού. Ε, δηλαδή λειτουργεί κάπως ως εντολοδόχος, ως προστάτης του λαού αυτού σημαίνει ότι ο κατέχον πρέπει να τηρεί τα ανθρώπινα και να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα του κατεχόμενου λαού, το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Πρέπει διαρκώς και μονίμως να προετοιμάζει το έδαφος για την επιστροφή των έδαφων, την επιστροφή της ε, ε, ανεξαρτησίας και την αρχή της αυτοδιάθεσης. Δεν μπορεί να έχει διάθεση αρπακτική, δεν μπορεί να λαφυραγωγεί ή να ε, ληστεύει και να Δεν μπορεί να γίνονται απελάσεις λόγου χάρη. Η μόνη εξαίρεση εδώ είναι ότι οι κατεχόμενοι και ο λαός των κατεχομένων και των κατεχόντων πρέπει να λειτουργούν με βάση, ως, με βάση την ασφάλεια, με αυτό ως βασικό τους γνώμονο. Και η τέταρτη αρχή σε σχέση με την κατοχή είναι ότι ο θα πρέπει να δρά εν καλή πίστη. Η καλή πίστη είναι ακρογωνίως λίθος του διεθνούς δικαίου. Η απέτηση περί καλής πίστης ε, βρίσκεται και στη χάρτα των, του ΟΗΕ, στη Σύμβαση της, Βιέννας, σε όλ, της Βιέννης, σε όλες τις διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες. Καλή πίστη σε σχέση με το κατεχόμενο. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές παράμετροι. Ο κατέχον που δικεί ένα κατεχόμενο, μια κατεχόμενη περιοχή θα πρέπει πρώτα απ' όλα να συμμορφώνεται με όλες τις ε, συστάσεις της διεθνούς κοινότητα, Δηλαδή ψηφίσματα που προέρχονται από την Γενική Συνέλευση, από το Συμβούλιο ασφαλεία, από το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο, από τα συμβαλώμενα μέρη στην ε, Σύμβαση της Γενέβη και έπειτα πρέπει να συμμορφούνται με όλα τις αρχές και τα συστατικά στοιχεία του διεθνούς ε, ε, δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτά όλα διέπουν, πρέπει να διέπουν τη συμπεριφορά του κατέχοντος. Ευτυχώς έχουμε ένα προηγούμενο εδώ μια από τις πιο γνωστές αποφάσεις στο διεθνές δίκαιο. 1971 απόφαση και συμβουλευτική ε, γνωμοδότηση από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την Αμίμπια. Εάν ε, σας πω σε 30 δευτερόλεπτα τι συνέβη από την πλευρά της ιστορίας η ε, Νότια Αφρική ως συντολιδόχος δύναμη ζήτησε εντολή από τον ΟΗΕ το 1982 για να δικήσουν την πρώην απικία της ιτημένης Γερμανίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου όλα αυτά τα εδάφη που ήταν πρώην απικίες θα γίνονταν μέρος ενός καταπιστεύματος του ΟΗΕ. Η Νότια Αφρική αρνήθηκε την ε, Δυτική Νότια Αφρική, δηλαδή την Αμίμπια, να την ε, ε, αφήσει να περάσει αυτό το καταπίστευμα. Ήσχε, λοιπόν εκεί και το Απαρτχάιντ και είχε ζητηθεί de facto προσάρτηση της Ναμίμπια. Η διεθνής κοινότητα το 1966, ενώ ήδη είχε αρχίσει να ανησυχεί, με τη Γενική Σύνελευση του ΙΕ δήλωσε ότι η εντολή η συνεχιζόμενη εντολή ε, της Νότιας Αφρικής επί της δυτική νότια Αφρικής, δηλαδή τη Ναμίμπια, ήταν πλέον παράνομη. Και μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1980, ε, το 1970 μάλλον, το Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε δύο ψηφίσματα, εκ των οποίων το δεύτερο επιβεβαίωνε ότι η συνεχιζόμενη διοίκηση της Νότιας Αφρικής επί της Ναμίμπια δεν ήταν πλέον νόμιμη. Και τον Ιούνιο του 1971 το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο έλαβε την απόφαση του και εξήβρε και επιβεβαίωσε τις περισσότερες από τις αρχές που ήδη είχαν εκφραστεί ε, και σας παρουσίασα εγώ εδώ μη προσάρτηση, ε, των καλύτερων συμφέρον του κατεχόμενου λαού και καλή πίστη. Τα, υπό τον καταπίστευμα αυτά εδάφη ήταν ε, υπό την ευθύνη της δύναμη κατοχή, που έπρεπε όμω να τα οδηγήσει στην κατάσταση τη αυτοδιάθεση και τη ανεξαρτησία. Και να μην γίνουν προσαρτημένα εδάφη με το πέρα του χρόνου. Αυτή η διαρκή παραβίαση των υποχρεώσεών τη από τη δύναμη κατοχή ε, έκανε την ε, συνέχιση της εντολής δίκησης αυτών των εδαφών παράνομη τελικά. Όλα αυτά, κατά τη δική μου την ε, εκτίμηση και την εισήγησή μου προς εσάς, ισχύουν ε, για την κατοχή του Ισραήλ, της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Αλλά και η εξουσία ε, εντολής και δίκησης που έχει το Ισραήλ δεν είναι πλέον νόμιμη. το πλαίσιο περί εντολοδόχου δυνάμεως συνεχίζει να ισχύει εφόσον εξυπηρετείται το ύψος των συμφέρων του κατεχόμενου λαού από την δύναμη κατοχής. Αυτά θέλω να ε, παρουσιάσω τη στιγμή που η Δυτική Νότια Αφρική προέκυψε από όσα ε, προέβλεπε το άρθρο 22. Και η πρόσφατη σύμβαση, η 40η σύμβαση, ε, η τέταρτη μάλλον σύμβαση ε, και το 22ο άρθρο είναι ε, παρακλάδια του ίδιου δέντρου στην ουσία. Ο αλλοδαπός κατέχων πρέπει να σέβεται το δικαίωμα των κατεχόμενων και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους. Η Συμβουλευτική Επιτροπή λοιπόν για την Ναμίμπια το 1971 βρήκε τρόπους ε, να κηρύξει παράνομη την κατοχή και αυτό είναι ένα προηγούμενο στο οποίο μπορούμε να κάνουμε διαρκή αναφορά και να παραπέμπουμε για την κατοχή των ε, Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ. Ε, και τώρα να περάσω στο ερώτημα κατά, για το κατά πόσον είναι παράνομη ένομη η κατοχή. Εάν ελέγξουμε τα κατά πόσον ισχύει κάθε μια από αυτές τις τέσσερις αρχές. Κατά πόσον παραβιάστηκε με τρόπο μόνιμο και συστηματικό από την αρχή κατοχής, τη δύναμη μάλλον κατοχή, νομίζω ότι εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για παραβιάσεις από τον κατέχοντα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι θεωρώ ότι στα 50 χρόνια κατοχής του Ισραήλ από την Παλαιστίνη, το Ισραήλ παραβίασε και τις τέσσερις από αυτές τις αρχές. Πρώτα απ' όλα σε σχέση με την προσάρτηση. Τον κανόνα περί μη προσάρτησης προσαρτήθηκε η Ανατολική Ιερουσαλήμ μέρη της Δυτικής Όχθης το 67 και το 80 και σήμερα το Ισραήλ έχει περάσει σε de facto προσάρτηση του μεγαλύτερου μέρους της ε, Λωρίδας της Γάζας. 60% περιοχή ΣΥ όπως ονομάζεται, με 60.000 Ισραηλινούς επικιστές και 225, 225 επικισμούς, σημεία επικισμού. Έπειτα, για το κατά πόσο είναι μόνιμη η προσωρινή κατοχή, σας εξήγησα ότι οι προσφατότερες ε, προσαρτήσει κατοχέ έχουν πολύ μικρότερη διάρκεια. Εδώ μιλάμε για 50 χρόνια σε σχέση με την ε, προστασία του ύψου του συμφέροντο του κατεχομένου λαού. Εδώ έχουμε μια κοινή γεωγραφική επικράτεια, μια κοινή γεωγραφική περιοχή, αλλά διαφορετικά δίκαια που ισχύουν, διαφορετικά πολιτικά δικαιώματα, διαφορετικά κοινωνικά δικαιώματα, οικονομικά και δικαιώματα πρόνοιας. Και όλα κρίνονται με βάση μία φυλή, μία εθνότητα. Υπάρχει λοιπόν πρόβλημα με την κοινωνική συνιστόσα και αυτό είναι παραβίαση των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με του νόμου που ε, ε, απαγορεύουν την διακριτική μεταχείριση. Και ενώ η οικονομία των Παλαιστινίων καταπιέζεται λόγω του διαμελισμού των ανταφών του, ε, είναι και αυτό παραβίαση του καλύτερου συμφέροντο, του του συμφέροντος του κατεχόμενου λαού από τον δύναμη κατοχή. Και η τέταρτη αρχή, η αρχή της καλής πίστης, ε, μπορώ να πω ότι το Ισραήλ δεν έχει σεβαστεί τι υποχρεώσει που προκύπτουν από τα άρθρα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, το Διεθνές Δίκαιο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, με τις διάφορες τιμωρίες που επιβάλλονται, με τη χρήση των φυσικών πόρων και ως προς την μη συμμόρφωση της επίβλεψη, της ε, τήρησης των αρχών της διεθνούς κοινότητας, το Ισραήλ δεν, παραβιά, δεν έχει σεβαστεί τουλάχιστον 40 πάνω από 40 ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και 160 ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τι θα πρέπει λοιπόν να συνάγουμε από όλα αυτά. Εγώ φρονώ ότι πρόκειται για ένα σοβαρότατο νομικό ζήτημα του διεθνούς δικαίου. Την μετατροπή ενός νόμου κατέχοντος που ε, εξελίσσεται σε παράνομο. Αλλά δεν είναι απλώς νομικό και νομικιστικό το ζήτημα εδώ. Γίνεται και πολιτικό φυσικά και διπλωματικό ταυτόχρονα. Το πλαίσιο απαιτεί νέα φιλοσοφία, νέα ε, επικοινωνία και διάδραση και νέα εργαλεία από τη διεθνή κοινότητα. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Θα πρέπει να ορίσουν την κατοχή ως παράνομη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να πάυσει η κατοχή και να οριστούν εθνικά και διεθνή δικαστήρια ώστε να εφαρμοστούν οι απαραίτητοι νόμοι να υπάρξει συνεργασία και να πάυσει η κατοχή. Η διεθνή κοινότητα ίσως θα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για να χρησιμοποιήσει ένα εύρωστο, νόμιμο ε, και αποτελεσματικό εργαλείο για να ε, υπάρξει συνεργασία με τις δυνάμεις κατοχής ε, και να υποχρεωθούν να πάψουν την κατοχή τους. Αυτό σας εισηγούμε σήμερα, ότι χρειάζεται να βρούμε ένα τρόπο για να κρίνουμε και άλλες ανάλογες κατοχές στον κόσμο. Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να σημειώσει ότι είναι διαρκής και συστηματική αυτή η κατοχή. Δεν θα πάψει από μόνη της. Δεν πρόκειται να τελειώσει, ούτε θα αντιστρέψει την πορεία της. Εκτός και αν υπάρξει μια δραματική αλλαγή στα διεθνή πράγματα ή το εσωτερικό status quo. Αυτό το πρέπει να λάβει υπόψη της η διεθνής κοινότητα και είναι απλώς ένα από τα πολλά εργαλεία που μπορεί να αντιστρέψουν την πορεία με άοκνες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών για να δοθεί τέρμα σε αυτή την κατοχή και να πάυσει ε, αυτή η εποχή κατοχής που θα οδηγήσει σε μια εποχή ελευθερίας και για τους Παλαιστινίους. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. για την πολύ εντυπωσιακή αυτή παρουσίαση για το μάθημα αυτό διεθνούς δικαίου, για την πολιτική και ηθική αξιολόγηση της κατοχής. Χρειαζόμαστε τέτοιου είδους μαθήματα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαλεντίνα Ζάροβα με, τα διδακτορική, ε, με τα διδακτορικό μέλος στο κέντρο παγκόσμιου δημοσίου δικαίου στο Πανεπιστήμιο Κότς της Κωνσταντινούπολης και νομική σύμβουλος του Δικτύου Παγκόσμιας Νομικής Δράσης. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, σας είμαι γνώμων που οργανώσατε αυτή την ε, εκδήλωση και που αφιερώνετε αυτό το χρόνο για να συζητήσετε μια έκθεση που ετοίμασα τον Ιούνιο του 2000... Συγγνώμη, τον Ιούνιο ε, του 2017, επευκαιρία της 50ης επαιτίου της κατοχής, με, όπου εξετάζουμε το ρόλο της ευθύνες για την κατάσταση, για ξένο έλεγχο που ασκεί το Ισραήλ στα Παλαιστινιακά εδάφη. Υπάρχουν άλλες έξι περιπτώσεις κατοχής ε, που είναι ατέρμονες. Με βάση τις ε, έρευνες που έχω κάνει επί χρόνια και με βάση τις ε, συζητήσεις που έχουν γίνει για την έκθεση αυτή από διεθνείς εμπειρογνώμονες, απεικονίζω κάποιες από αυτές τις σκέψεις στην έκθεση μου, είναι στη διάθεσή σας δημόσια, και εγώ θα σας κάνω τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, για το διεθνές νομικό πλαίσιο. Οι κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ δραστήριες ε, στα παλαιστινιακά κατεχόμενα εδάφη ε, για μια παράνομη και παρατεταμένη κατοχή. Ε, συγχαίρω τον κύριο Λίνξ για, για τα όσα είπε σχετικά. Δεύτερον, για το χαρακτήρα και τις επιπτώσεις των παράνομων δράσεων της Ισραηλινής κυβέρνησης και τέλος μια, ένα σύντομο προβληματισμό ε, πάνω σε αυτή τη δράση και για το τι πρέπει να κάνουν οι τρίτοι, ε, τα τρίτα μέρη ε, με βάση το διεθνές δίκαιο. Η έκθεση ξεκινάει με ένα απλό ερώτημα. Ποιες είναι οι συνέπειες ε, του διεθνούς δικαίου σε περίπτωση που υπάρχει ξένος εδαφικός έλεγχος ή κατοχή που συνεχίζεται και διατηρείται δια της βίας με σκοπό να προσαρτηθούν μονίμως τα εδάφη ή να μετασχηματιστούν να μετασχηματιστεί το διεθνές καθεστώς των εδαφών αυτό μονίμως. Προσπαθούμε να καταλάβουμε τις συνέπειες ε, και να δώσουμε απαντήσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό έχουμε μία προσέγγιση επίτηδες ε, συντηρητική για το τι λέει το διεθνές ε, δίκαιο. ο όρος ε, παράνομος και παρατεταμένος, ε, παράνομη και κατεταμένη κατοχή προσπαθεί να απεικονίσει το, τη ζημία που γίνεται ε, πάνω σε κάποιους με τη χρήση βίας, απειλής για να παραταθεί μια κατάσταση κατοχής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις Έχουμε την παρουσία των δυνάμεων κατοχής ε, στα κατεχόμενα εδάφη που δημιουργούν μια παράνομη κατάσταση που παραβιάζει ουσιαστικά την απαγόρευση για την απόκτηση εδαφών δια της βίας, άρθρο 24 ε, της ε, χάρτας του ΟΗΕ, του εθνικού δικαίου και που θεωρείται ως κανόνας του διεθνούς δικαίου από όλους. σε ορισμένε περιπτώσει ε, πολλά κράτη θεωρούν ότι αυτέ οι δράσει ε, αποτελούν μορφή βία. Τρει επιπτώσει τη ε, κατοχή απεικονίζουν αυτή την πραγματικότητα της παράνομης παρατεταμένης κατοχής που συζητάμε στην έκθεση. Καταρχά μία κατοχή που επιβεβαιώνει την de jure ή de facto προσάρτηση όπως η κατοχή του Ισραήλ ε, των Παλαιστινιακών εδαφών, ε, η κατοχή της Κρυμαίας από τις ρωσικές δυνάμεις και αυτή είναι περίπτωση κατοχής, η παράνομη ε, προσάρτηση και διαχείριση της Δυτικής Σαχάρας από το Μαρόκο. Άλλη περίπτωση. Μια δεύτερη κατηγορία τέτοιων περιπτώσεων είναι σε περίπτωση που υπάρχει μόνιμος εκτοπισμός κατοίκων και μόνιμη κατοχή τμήματος της, ε, των εδαφών αυτών. Ε, με σκοπό να οδηγηθούμε σε, σε απόσχεση ενός τμήματος του κάποιων εδαφών. Παραδείγματο χάρη στην Τουρκία, στην, ε, όπως κάνει η Τουρκία στην Κύπρο. Ρωσία στην υπερνηστερία, ε, στην Γεωργία και στην ε, Νότια Οσετία. Το Αζερβαϊζάν στο Ναγόρνο Καραμπάν. Όλες αυτές οι κατοχές ε, είναι ίσες. Ε, στα μάτια του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ε, στα πλαίσια του δικαίου για την ε, διαχείριση των περιοχών συγκρούσεων. Δεν υπάρχουν καθόλου σε καμία περίπτωση λόγοι κατοχής. Το να υπάρξει διαμεσολάβηση σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι, σε αυτά τα εδάφη που είναι υποκατοχή, δεν μπορεί να... δεν είναι μια εύκολη λύση. γιατί ε, η διαμεσολάβηση ακριβώς, ε, ακριβώς θέλει να ακυρώσει τις ε, προσπάθειες των δυνάμεων κατοχής. η κατοχή στην πραγματικότητα δημιουργεί μια κανονιστική μετατροπή στο διεθνές δίκαιο. Μια αλλαγή από διαχείριση μιας σύγκρουσης ε, σε πρόληψη της, σε πρόληψη της σύγκρουσης. Αυτά είναι στοιχεία του δικαίου που διέπουν τις περιοχές ε, συγκρούσεων. Ε, και θα πρέπει να προσαρμοσ... να γίνουν κάποιες προσαρμογές στο διεθνές δίκαιο. Το σωστό νομικό πλαίσιο που αναφέρει η έκθεση είναι μια ενσωματωμένη προσέγγιση που θεωρεί ότι πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η αρχή της απαγόρευσης της βίας ε, με βάση το διεθνές δίκαιο. Μια αντίστοιχη περίπτωση είναι η αλληλεπίδραση διεθνούς ε, ανθρωπιστικού δικαίου και διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το διεθνές δίκαιο ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα συμπληρώνει και εφαρμόζεται παράλληλα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Αλλά σε περίπτωση κατοχής ε, πρέπει να, γίνεται σεβασμό, να υπάρχει σεβασμός του ανθρωπιστικού ε, δικαίου και να σταματήσουν να συμβαίνουν οι δημογραφικές αλλαγές στα κατεχόμενα εδάφη που στρεβλώνουν την προστασία των δικαιωμάτων ε, στα εδάφη αυτά από τις ε, δυνάμεις κατοχής ή από το κράτος κατοχής. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι συνέπειες αυτής της αλλαγής στο νομικό πλαίσιο είναι τριπλές. Καταρχάς η παρουσία του, των δυνάμεων κατοχής στα κατεχόμενα εδάφη είναι παράνομη και θα πρέπει πάρα αυτά να σταματήσει. Τον, υπάρχει υποχρέωση απόσυρσης από, στις δυνάμεις κατοχής, αλλά υποχρέωση και για τη διεθνή κοινότητα και τα τρίτ, ε, τις τρίτες χώρες και τους διεθνείς φορείς. Επίσης, ε, οι διοικητικέ πράξει των δυνάμεων κατοχή ακυρώνονται από το διεθνέ δίκαιο. Φυσικά υπάρχουν όρια ε, στην ακύρωση των διατάξεων των δυνάμεων κατοχή ή του κράτου κατοχή, ε, αλλά λόγω τη χρήση βία θεωρείται παράνομη οποιαδήποτε πράξη και δεν μπορεί να αναγνωριστεί και να εφαρμοστεί από τρίτα μέρη. Αυτό συμπεριλαμβάνουν φυσικά την ε, παράνομη αναθεώρηση της πολιτικής και οικονομικής τάξης, αλλά και το δικαίωμα και την περίπτωση ας αλλαγής του διοκτησιακού καθεστώτος ε, ε, και παράνομες ας πούμε, οικονομικές ροές που συμπεριλαμβάνουν και μέρη εκτός αυτών των εδαφών. Δηλαδή συναλλαγές και πράξεις ανάμεσα σε άτομα των εδαφών αυτών και άτομα που ζουν εκτός. Υπάρχουν κάποια όρια που θέτει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Στην περίπτωση του Ισραήλ, μέσω του πλαισίου αυτού και των συνεπειών, βλέπουμε τις ε, ιδιαίτερες δραστηριότητες και πολιτικές που προωθούνται στα κατεχόμενα και υπό το Διεθνές Δίκαιο και σε ό,τι αφορά την, ε, τον τρόπο που, ασκεί το Διεθνές Δίκαιο το Ισραήλ και τα προβλήματα που δημιουργεί. Κυρίως η κατοχή της ε, δυτικής όχθης από το Ισραήλ ε, θεωρείται ε, παράνομη προσάρτηση του μεγαλύτερου μέρους του εδάφους αυτού. Δεν χρειάζεται η προσάρτηση να γίνει μέσω επίσημης πράξης, αρκεί ο επίσημος έλεγχος του εδάφους αυτού, ουσιαστικός μάλλον έλεγχος του εδάφους αυτού, και προκύπτει από ένα μακρύ κατάλογο μέτρων, για την αναθεώρηση ας πούμε της, ε, του, νόμι, του καθεστώτος ε, που διέπει τους επίκους, ε, το δικαίωμα διαμονής στα κατεχόμενα εδάφια από Ισραηλινούς κτλ. Επίσης, κανονικά δεν θα πρέπει να γίνεται δεν γίνεται μάλλον διαχωρισμός ανάμεσα σε παλαιστινιακά εδάφη και σε ε, Ισραηλινά εδάφη με βάση την ε, εσωτερική Ισραηλινή ένωμη τάξη. Επίσης, η, η στάση της Ιταλιανής κυβέρνησης ε, από τις... τα πρώτα χρόνια της κατοχής μέχρι σήμερα δείχνει ακριβώς τα προβλήματα. Φυσικά αυτά δεν είναι καινούρια στοιχεία, ε, αυτές οι νομικές διατάξεις, αλλά δεν είναι, είναι σημαντικά για να καταλάβουμε τι μπορεί να πει, ε, τι απαντήσεις μπορεί να δώσει το διεθνές δίκαιο. Και γενικά ε, το συμπέρασμα είναι ότι η κατοχή ήταν επιζήμια. Φυσικά θα πρέπει να σταματήσει η χρήση βίας Αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω διεθνούς διατησίας. Συχνά μπορεί να γίνει και σε επίπεδο τρίτων μερών, μεμονωμένων κρατών ή και με μεμονωμένων φορέων ε, διασυνοριακών, ας πούμε, ή υπερεθνικών, ας πούμε, εταιριών. Οι διεθνείς αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς έχουν ε, το δικαίωμα να, και την υποχρέωση να θέσουν τέρμα στο καθεστώς αυτό. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν και οι απαραίτητοι μηχανισμοί ούτως ώστε να διευκολυνθεί μία αναγνώριση του καθεστώτος αυτού. Θα πρέπει, τελειώνοντας, να σας πω ότι ο σκοπός αυτής της ανάλυσης στην έκθεση δεν ήταν να αξιολογήσουμε είτε τη δέσμευση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των τρίτων Κροτών ε, απέναντι στα, τρίτα, απέναντι στα μέτρα αυτά, παρότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Το θέμα είναι να πούμε στους ε, πολιτικούς, στους δικηγόρους και σε όλους τους ενδιαφερόμενους ποιο είναι το, το πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε και ο καθηγητής Λίνκ για να αντιμετωπιστούν αυτές οι παράνομες καταστάσεις όπως αυτή της ε, Ισραηλινής κατοχής. Και για να προωθηθεί διαδικασία μία αναγνώρισης με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό το πράγμα δεν έχει προωθηθεί μέσω άλλων διαδικασιών σε διεθνές επίπεδο. Και για να υποστηριχθούν ε, προσπάθειες για να γενικευθεί αυτή η αντιμετώπιση πέρα από την περίπτωση της κατοχής του Ισραήλ, από το Ισραήλ της Παλαιστίνης. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε που αναπτύξατε το θέμα της κατοχής εξηγώντα ότι δεν υπάρχουν καλές και κακές κατοχές ούτε Παραδεκτέ ή απαράδειε κατοχέ βάσει του κοινωνικαίου. Και ότι θα πρέπει να αποσχούμε από υποκριτικέ τοποθετήσει όπου μερικέ από τι κατοχέ είναι καλύτερε από άλλε. Η απαραδεκτε κατοχε είναι δικαιου και είναι απαράδεκτη. Τέρμα στις κατοχές. Αυτό τις κατοχε το γενικό συμπέρασμα όσων είπατε. Και ειναι απαραδεκτη τερμα στις κατοχε αυτο ειναι το γενικο συμπερασμα οσων ειπατε και τωρα να στραφώ στον κύριο Χάμερμπεργκ. Και να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν ειδικό απεσταλμένο του Συμβουλίου της Ευρώπης και Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και βεβαίως σας ξέρω από πολλά χρόνια γιατί βρίσκεται πρέσβη στη χώρα μου της Σουηδίας. Παρακαλώ κύριε Χάμερμπεργκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Να πω καταρχάς ότι στηρίζω πλήρως τα σχόλια της ε, Βαλεντίνα και το νέο βλέμμα που την ακατεύθυνση που έδωσε στη συζήτηση. Νομίζω ότι το έγγραφο και το όσο μας παρουσίασε ο Μέγλινγκ είναι ε, ύψης της σημασίας. Ελπίζω να ε, λάβουν γνώση όσο το δυνατόν περισσότερο και να συζητηθούν ευρέως όχι μόνο στις δομές των ΗΠΑ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παντού. Είναι βασικά ζητήματα αυτά τα οποία αναπτύσσονται και πολλά βρέθηκαν στη σκιά της προπαγάνδας και άλλων προσπάθειων να υπονομεύσουν την όλη προσπάθεια για την ειρήνη και τη συζήτηση και να δούμε το τι ακριβώς σημαίνει κατοχή. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο θα γίνει αντιληπτό σε ένα έγγραφο ιδιαίτερα εξειδικευμένο για να φωτίσει την όλη συζήτηση του θέματος που μας απασχολεί. Προσάρτηση λοιπόν, να ένα θέμα που μας απασχόλησε πολύ ως τώρα και μετά τον πόλεμο το 1967 προσαρτήθηκε η Ιερουσαλήμ. Αυτό που βλέπουμε όμως σήμερα είναι ότι όχι απλώς συνεχίζεται αυτή η τάση, αλλά έχει μάλιστα αυξητική Τάση η προσάρτηση σε σχέση με το παρελθόν. Αυτά που συζητιούνται στην ΚΝΕΣΕ τώρα είναι το αν θα υπάρξει πολύ ε, ευρύτερη προσπάθεια προσάρτησης της περιοχής ΣΥ όπως έχει ονομαστεί αυτό βρίσκεται στο φως των προβολέων όταν μιλάμε για προσάρτηση, αλλά μπορεί να πάνε τα πράγματα ακόμη μακρύτερα. Η συζήτηση λοιπόν έχει ξεφύγει από την κλασική έννοια της κατοχής μετά τον πόλεμο, όπου ο κατέχον έμενε στο κατεχόμενο έδαφο για κάποιο διάστημα, όχι πάρα πολύ, για να προστατεύσει υποτίθεται τα συμφέροντα του κατεχόμενου πληθυσμού και μετά ε, μπορούσε να παραδώσει την εξουσία σε ένα άλλο καθεστώ, μια άλλη κυβέρνηση που θα προστατεύει αυτό το λαό από μια καινούργια θέση. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Έχουμε μετακινηθεί προς την ε, προσάρτηση, η οποία φαίνεται να είναι πλέον ε, ολοκληρωμένη σε ό,τι αφορά τα εδάφη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να περάσει ως μήνυμα. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να τονίσουμε και στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση είναι η απόκριση της Ισραηλινής κυβέρνησης στα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ασφαλείας το 23-34. Όχι απλώς ε, η λεκτική απάντηση στο ψήφισμα έλειψε, αλλά υπήρξε μια εντατικοποίηση της λήψης αποφάσεων για επικισμούς και για την προσάρτηση. Αυτή ήταν η απάντηση στην απόφαση, η οποία ε, ελήφθη σχεδόν ομόφωνα. Δεν την καταψήφισε κανείς. 14 ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος και μία χώρα, είπα ΕΠΑ, απήχαν. Η ύψιστη αρχή ερμηνείας του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, λοιπόν, και του διεθνούς δικαίου γενικότερα στον τομέα αυτό, ε, δεν έλαβε καμία απάντηση. Ίσα ίσα πήγαν ενάντια σε όσα ήθελε το Συμβούλιο Ασφαλείας να παρεμποδίσει και έλαβαν ακόμη περισσότερες αποφάσεις οι Ισραηλινοί. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επικεντρωθώ όχι τόσο πολύ στην νομική διάσταση του ζητήματος, που ούτως ή άλλως μας αποσχολεί εδώ, αλλά λίγο περισσότερο σε αυτό που ανέπτυξε ο Μάικλ Λίνκ και το όρισε ως καλύτερο ύψιστο συμφέρον του κατεχομένου λαού και καλή πίστη. Δηλαδή το κατά πόσο ο κατέχον πρέπει να αποσχολείται με τον λαό που κατοικεί σε μια κατεχόμενη περιοχή. Είναι πολλά αυτά που θα είχα να πω εδώ. Το γεγονό ότι οι επικισμοί εντάθηκαν είναι γεγονό, αλλά μα απασχολεί την καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων στι κατεχόμενε περιοχέ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τι έγινε σε ό,τι αφορά την ίδρυυση, την πρόσβαση στο νερό. Θα έλεγα ότι ήδη εδώ βλέπουμε μια πολιτική κλοπή σε ό,τι αφορά το νερό. Το νερό σε αυτή την περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Το ότι το ε, λαιλατούν και το χρησιμοποιούν οι κατέχοντες με παράδειγμα τρόπο είναι χαρακτηριστικό. Οι δρόμοι που χτίστηκαν. Μερικοί από τους δρόμους αυτούς είναι μόνο για τους κατέχοντες, τους επικιστές και όχι για τους Παλαιστινίους. Αυτό έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των ανθρώπων στην περιοχή αυτή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο η οικοδόμηση του τείχους διαχωρισμού. Και αυτό είχε μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την ε, καθημερινότητα, τα προβλήματα στέγασης πολλών Παλαιστινίων σε αυτή την περιοχή. Εγώ ενδιαφέρθηκα όλος ιδιαιτέρως για το πώς ζουν τα παιδιά στις κατεχόμενες περιοχές και για ένα διάστημα πριν από πολλά χρόνια είχα αναλάβει με εντολή της καναδικής κυβέρνησης η οποία ήταν επικεφαλής σε σοβαρές προσπάθειες να συζητήσουμε την κατάσταση των παιδιών, των προσφύγων, των, των προβλημάτων των προσφύγων γενικότερα. Εκεί λοιπόν είχα αναλάβει ως ειδικό απεσταλμένο για τα παιδιά στους καταβλημούς των προσφύγων στην Δυτική Όχη και στη Γάζα και προσπάθησα να ε, αναπτύξω ε, δράση για όλα τα παιδιά των Παλαιστινίων Έκτοτε, όσε φορέ επέστρεψα στην περιοχή, είδα ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Έχει με κατά πολύ. Παιδιά που έζησαν συνθήκε πολέμου, πολύ δυσάρεστε, φυσικά και είχαν επιπτώσει στην ψυχολογική του υγεία, ε, τραυματικέ εμπειρίε και ένα από τα βασικά προβλήματα των οικογενειών εκεί είναι η κακή ψυχολογική για των παιδιών. Το τραύμα είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις ζωές των παιδιών αυτών και βεβαίως έχει να κάνει με την ε, κατοχή. Εάν κανείς απαριθμίσει όλες τις διαφορετικές πτυχές που ε, σχολιάστηκαν εδώ, δεν μπορεί να φτάσει παρά μόνο σε ένα συμπέρασμα. Ότι η κατοχή πρέπει να πάυσει. Είναι παράνομη και θυματοποιεί, φέρνει στη θέση του θύματο ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του σε μεγάλη κλίμακα, η οποία δεν θα μπορούσε να είναι αποδεκτή. Και επίση πρέπει να διεξάγουμε το συμπέρασμα ότι δυστυχώ η πολιτική αυτή υπονομεύει μακροπρόθεσμα την εξέβρεση ειρηνική λύση. Όσο περισσότερο τραβάει αυτή η κατάσταση κατοχή, τόσο πιο απίθανο γίνεται να βρεθεί λύση λύση ειρήνη στις συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών. Δυσκολεύεται το έργο για την ειρήνη. Είναι κάποιοι που θα έλεγαν ε, ότι εμείς ε, και πολλοί από όσους συμμετέχουμε εδώ στο πάνελ, όπως ο Μάικλ Λίνξ, είμαστε κατά του Ισραήλ. Όχι. Θα πρέπει τους Ισραηλινούς να του πάρουμε σοβαρά, αλλά και οι ίδιοι να αναλάβουν ευθύνε για να σκεφτούν τι κάνουν οι ρετοί εκπρόσωποι του, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του, στο όνομά του. Στο Ισραήλ δεν μπορούμε να παραπευθύνουμε επικριτικά σχόλια, καθώ υπάρχουν και συστηματικέ παραβιέσει του διεθνού ε, ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνού δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορούμε να εντυπωσιαζόμαστε από τι διαδικασίε προπαγάνδας και να αφαιθούμε στις προσπάθειες να παρεμποδιστούν οι συζητήσεις για τα θέματα αυτά. Γι' αυτό θεωρώ τόσο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, λάβει στάση ε, ενεργό στην όλη κατάσταση, να προσπαθήσει να ορίσει ως παράνομη την κατοχή και να συμβάλλει και στις όλες συζητήσεις των ΟΗΕ να ασχοληθεί με την διεύθυνση των ε, καλύτερων δυνατών διμερών σχέσεων και γι' αυτό σας εύχομαι καλή τύχη σε αυτές τις προσπάθειες. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ, κύριε Χάμερμπεργκ. Τονίσατε το στόχο της σημερινής συζήτησης. Να προωθήσουμε κάποιες δράσεις με ομοφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτως ώστε να σταματήσουμε καταρχήν την κατοχή και να δώσουμε τη δυνατότητα στους Παλαιστίνιους να ζήσουν με ασφάλεια και ειρήνη και να οικοδομήσουν τη χώρα τους. Τώρα, για 10 λεπτά θα ακούσουμε ερωτήσεις και θα δοθούν απαντήσεις. Θα ήθελα να δώσω το λόγο, ε, το λόγο καταρχάς στην κυρία, στον κύριο Μαχτά και ε, συνεχεία στην κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είμαι πιο σύντομο από τα 10 λεπτά. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση στον κύριο Πρέσβη τον, το, και τον ειδικό απεσταλμένο του κυρίου Αμπάς. Αν θα έχουμε την ευκαιρία. Ακούσαμε δύο ειδικού από το Διεθνές Δίκαιο. Πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Μιλήσατε για όλες τις εκθέσει, όλα όσα παραβιάζει επί χρόνια το Ισραήλ. Επομένω, το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί. Γιατί το Ισραήλ έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που κάνει. Φυσικά η απάντηση είναι προφανή όσο και η ερώτηση. Γιατί κανεί δεν κάνει τίποτα άλλο. Τίποτα. Και το ερώτημα που τίθεται εν συνεχεία είναι, μα γιατί δεν κάνει κάποιο κάτι. Εδώ, εδώ και τρία χρόνια εγώ είμαι ευρωβουλευτή. Ε, δεν, έχω, δεν είμαι υπέρμαχος των Παλαιστίνιων, ε, δεν τους υπερασπίζουμε. Ε, μάλιστα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι ίδιοι Παλαιστίνοι κτλ. Ε, στη χώρα μου μάλιστα έχω το στίγμα του, του προπαγανδιστή των, υπέρ των Παλαιστίνιων και του αντισημίτη. Τι μπορούμε να περιμένουμε από την πολιτική των δύο κρατών. Ε, στο, στον ΟΗΕ ψηφίζονται συνεχώ ε, ψηφίσματα. Και εμεί ψηφίσαμε ένα ψήφισμα. Ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το κράτο τη Παλαιστίνης, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το ερώτημα είναι λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε από τι πολιτικέ. Δεν θα έπρεπε καταρχά να στραφούμε προ την κοινωνία των πολιτών, να την πιέσουμε, ή μάλλον να πιέσουμε μέσω τη κοινωνία των πολιτών. Και μπορεί να κάνω και μια βλακώδη ερώτηση, αλλά θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Εγώ ως πολίτης, η κοινωνία των πολιτών, μπορώ να απευθυνθώ στα διεθνή δικαστήρια και να ε, ισχυριστώ ότι δεν υπάρχει σεβασμός διαφόρων ψηφισμάτων. Γιατί αν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Από τον Ιανουάριο του 2018 θα έχουμε όλοι μπει σε προεκλογική εκστρατεία. Ο κύριος ε, Γιούνκερ, ο κύριος Μακχό ε, ετοιμάζουν ήδη τις εκλογές, τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2019. Ίσως Μήπως θα έπρεπε ο κύριος Μαχμούτα Αμπάς να κάνει το γύρο των ευρωπαϊκών πρωτευουσών ούτω ώστε να συζητείτε το θέμα των Παλαιστίνιων και προεκλογικά πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές. Σας ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο, αυτά τα όσα, για τα όσα είπατε που ήταν περισσότερο σχόλιο παρά ερώτηση. Ας απαντήσουν οι ομιλητές του πάνελ. Κύριε Χάμερμπεργκ, θέλετε να πάρετε το λόγο να απαντήσετε. Το θέμα της αναγνώρισης της ε, Παλαιστίνης είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα. Γιατί μόνο όταν υπάρξει έναν εξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος θα υπάρχει δυνατότητα διαπραγματεύσεων ε, επίσης όρις με τους Ισραηλινούς. Η έλλειψη αναγνώρισης είναι πρόβλημα σήμερα. Υπάρχει μια έλλειψη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει συστήσει την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Και διάφορες κυβερνήσεις ε, που τις προσεγγίσαμε ε, δεν το έχουν κάνει. Η Σουηδία αναγνώρισε την Παλαιστίνη ως κράτος πριν από τρία χρόνια. Και υπήρχε τότε η ελπίδα στη Σουηδία θα ακολουθήσουν διάφορες άλλες ε, χώρες. διάφορα κοινοβούλια συνέστησαν στις κυβερνήσεις τους να το κάνουν. Αλλά οι κυβερνήσεις αγνόησαν τη σύσταση των δικών τους κοινοβουλίων. Γιατί? Λόγω της πίεσης από, το, από τη Ουάσιγκτον, ε, πίεσης από τους Ισραηλινούς. Αποφάσισαν δεν θέλουν να μπουν στον κόπο. Εγώ νομίζω ότι είναι και καινή ώρα για να τονίσουμε τη σημασία ε, που θα έχει η επίλυση αυτής της σύγκρουσης. Και δεν πρόκειται να επιληθεί εάν δεν δώσουμε προτεραιότητα στην, στο θέμα αυτό της πίεσης. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση ε, να υπάρξει σεβασμός του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Πίεση. Πίεση. Πιέστε λοιπόν, κύριε Λίνκ. Όλες οι παρατηρήσεις του κυρίου Μαχτά είναι πολύ έξυπνε. Ε, μίλησε για την ε, διεθνή νομική αποδοχή. δεν ε, η αδράνεια δεν είναι αποδεκτή. Δεν μπορεί κάθε, ε, οι χώρε, πούμε, να ξέρονται από πράγματα που ισχύουν για όλου του άλλου. Το άρθρο 25 λέει ότι τα μέλη του ΟΗΕ δέχονται ε, την ε, εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας με βάση την χάρτα αυτή. Το πιο πρόσφατο ψήφισμα, όταν υιοθετήθηκε, το Δεκέμβριο του 2016 14 ψήφοι κατά και μία αποχή. Αμέσως μετά από αυτό ο Πρωθυπουργό του Ισραήλ θεώρησε ότι είναι παλαβό αυτό το ψήφισμα. Δεν ε, είχαν κανένα σκοπό να σεβαστούν τις υποχρεώσεις που έχουν όλα τα μέλη του ΟΗΕ να δεχτούν τα ψηφίσματα. Κοιτάξτε, μιλήσατε για κάτι που απελπίζει όλους όσους ασχολούνται με το διεθνές δίκαιο. Ε, το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται από μόνο του. Ε, αυτό το αναγνωρίζει και το Διεθνές Δικαστήριο στην απόφαση του 1971 για την Αμίμπια, όπου είπε ότι το να χαρακτηριστεί μια κατάσταση σαν παράνομη δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει αυτή η παρανομία. Είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα ούτω ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση, το να γνωστεί ω παράνομη. Ελπίζω ότι τα δικά μου επιχειρήματα και η δική μου έκθεση, ότι αν θεωρήσουμε ότι είναι παράνομη δύναμη κατοχή στο Ισραήλ, τότε θα δημιουργήσει μια χιονοστιβάδα που θα μας οδηγήσει σε ένα τέλος. Το να θεωρήσει το Διεθνές Δικαστήριο ε, ότι υπάρχει μια παρανομία και η Γενική Συνέλευση Όπω ακριβώ συνέβη με την γνωμοδότηση αυτή για την Αμίμπια. Μαζί με μια σταθερή ε, πίεση της διεθνούς κοινότητας ε, απέναντι στις δυνάμει κατοχής, μπορεί να βοηθήσει ε, στην ελευθερία των Παλαιστινίων και στην πάυση της κατοχής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να χυθεί περισσότερο αίμα και με το να παρετηθούμε εντελώ, ας πούμε, ε, από το, ε, το διεθνές δίκαιο. Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πράγμα που μας ενώνει. Ε, η, θρησκεία μας, μας χωρίζει, η φυλή μας χωρίζει, η ιδεολογία μας χωρίζει, τα πάντα, η θρησκεία. ενώ εκεί υπάρχουν όλες οι αρχές που τις σεβόμαστε όλοι για το πώς θα μεταχειριζόμαστε οι τους δε. Γιατί αν αγνοήσουμε το διεθνές δίκαιο τότε πραγματικά φτύνουμε στο πιάτο μας. Επίσης, ε, το διεθνές δίκαιο δεν προστατεύει μόνο το κοινό συμφέρον και τους κανόνες, τους κοινούς διεθνείς κανόνες που δημιουργούν και ένα αξιακό σύστημα και που είναι απαραίτητο για τη ζωή μεταξύ κρατών και για την ε, ειρήνη και την ασφάλεια. Ε, συνδέεται και με την εσωτερική ένωμη τάξη. Αυτό το συνειδητοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, από το 2012 δημόσια με διάφορες θέσεις ε, που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ε, μέσω των συμπερασμάτων του ε, ε Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, Εξωτερικών Υποθέσεων. Και με βάση το 2334 στην παράγραφο 4 θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα ούτω ώστε να διακρίνουμε ανάμεσα στα Παλαιστινιακά και στα Ισραηλινά εδάφη. Ε, η μία αναγνώριση ε, προκύπτει από την ε, ακύρωση και την, τον, της νομιμότητας των επικισμών. Και το διεθνές δίκαιο είναι υπερισχύει της εσωτερικής ένομης τάξης. Δεν θέλω να μπω σε πιο πολλές λεπτομέρειες για τις ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ισραήλ. Ε, νομίζω ότι αυτό θα συζητηθεί στο δεύτερο πάνελ. Αλλά από τη σκοπιά του διεθνούς ε, δικαίου, αυτή η σχέση ανάμεσα στο διεθνές ε, δίκαιο και στην εσωτερική τάξη είναι πολύ σημαντική. Και το βασικό είναι ε, η μη αναγνώριση όλων αυτών των ε, κινήσεων, ε, των επικισμών κτλ. Γίνεται αυτό, αλλά γίνεται πολύ αργά. Και γίνεται λοιπόν με βήματα πολύ αργά και με νομικά κατασκευάσματα που είναι πολύ άκαμπτα. Ελπίζω και άλλα κράτη να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάργκρετ Άουγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις εξαιρετικές σας παρουσιώσεις. Εγώ πάσχω από το MDS, το Σύνδρομο Κατάθλιψης Μέσης Ανατολής. Μόλις σκεφτώ την παράνομη κατοχή, αμέσως το παθαίνω. Παθαίνω κατάθλιψη. Παρ' όλα αυτά, ήθελα να θέσω κάποιες ερωτήσεις και προς τους τρεις σας προς τον κύριο Λίνκ. Από όσα άκουσα να λέτε, έχετε πάει μακρύτερα από ότι εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο. Είπατε ότι η στρατηγική διαφοροποίηση είναι αυτή που πρέπει να εγκρίνουμε. Και κάθε φορά που το Ισραήλ μας κατηγορεί ότι χρησιμοποιούμε όρους όπως κατοχή, θα πρέπει να τα σπρώξουμε όλα σε αυτό το καλάθι, αλλά ε, ανοίξαμε το δρόμο προς αυτό το καλάθι λέγοντας ότι είναι παράνομη η κατοχή. Δηλαδή δεν πρέπει απλώς να γίνει διαφοροποίηση, πρέπει να ασκήσουμε πίεση στο Ισραήλ. Και θα πρέπει να κάνω και μια-δυο σκέψη παρατηρήσεις εδώ. Ξέρετε ότι το Ισραήλ μας απαγορεύει από το 2011 να πάμε στη Λουρδά της Γάζας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώς δέχεται το δέχεται. Το κοινοβούλιο, η προεδρία του κοινοβουλίου το δέχεται. Και αυτό διαρκεί. Διαρκεί σε τιμωρησία είναι αυτή. Και αυτό είναι πολύ επικίνδυνο για τις δύο πλευρές. Απλώς ήθελα να μου πείτε αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο, να πιέσουμε περισσότερο με ό,τι μεση διαθέτουμε για κυρώσεις Και επίσης να ευχαριστήσω τη Βαλεντίνα για τον τρόπο που ανέφερε και άλλες κατοχές οι οποίες τείνουν να λησμονηθούν. Πρέπει να το πάρουμε σοβαρά όλο αυτό το θέμα. Είπατε ότι υπάρχει ένας κατάλογος κατοχών που θα πρέπει να δουν και μια σειρά από συνέπειες θα πρέπει να δουν οι Ευρωπαίοι πολιτική. Και υπάρχει μια σειρά από συνέπειες για τις επιχειρήσεις. Εδώ νομίζω ότι είναι λίγο αβάσιμο το επιχείρημα ότι η κατοχή είναι παράνομη, ένομη και ούτω καθεξής. Διαρκώς με τον τρόπο αυτό, αυτό που λέμε στους Παλαιστινίους θα πάρετε τα ψίχουλα ό,τι και αν γίνει. Ό,τι λύση και αν βρεθεί. Ακούσαμε το 22% της ιστορικής Παλαιστίνης. Αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό αν σκεφτούμε ότι θα δημιουργηθεί κράτης, κράτος. Και θα πρέπει να προσέξουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε. De facto προσάρτηση και ούτω καθεξής. Διότι είναι σαν να λέμε σε όλους ότι μπορούμε να παραδώσουμε τα όπλα και να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών. Αλλά αν δείτε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο σήμερα, δύο κράτη, δείτε τι έγινε με την Ιουγκοσλαβία. Για μένα ένα κράτος ήταν εκρηκτικό ως λύση. Πρέπει να παραμένουμε πιστοί στη μόνη δυνατή λύση Δείτε τι έγινε μετά τις ε, σταυροφορίες. 200 χρόνια παρουσία στην περιοχή διατήρησαν. Ε, δεν λέω τώρα ότι θα πρέπει να γίνουν όλοι φίλοι εκεί αν θέλουν να διατηρήσουν την παρουσία τους. Πάντω και πάλι σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σα. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο εσεί κύριε Λίγκ. Ναι, και καταλαβαίνω δεν έχουμε και πολύ χρόνο, οπότε θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα. Οι ερωτήσει σα ήταν πολύ καλέ. Θα απαντήσω ω εξή. Ναι, προσπαθούμε να, να χαρακτηρίσουμε παράνομη την κατοχή του Ισραήλ. Ε, δηλαδή να πούμε ότι δεν υπάρχει νομιμοποίηση στην κατοχή. ε, οποιοδήποτε προσπαθεί να κάνει διάκριση μεταξύ των δύο θα πρέπει να έχει μια σαφή απάντηση. Ω προ την δύναμη που έχει η Ευρώπη, το Ισραήλ είναι ένα κράτος εμπορευόμενο. Ε, βασίζεται στους εμπορικούς του εταίρους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα πολύ σημαντικό εμπορικός εταίρος. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι εδώ έχετε κάποια δυνατότητα άσκησης πίεσης και αν ακούσετε προσεκτικά Του Ισραηλινούς που έχουν κάποια συνείδηση και είναι και γνωστέ προσωπικότητε. Ο αρχισυντάκτης της ε, βασικής εφημερίδα του Ισραήλ λέει σε σχέση με την κυβέρνηση της χώρα του ότι η διεθνής πίεση είναι ακριβώ το είδο δύναμη που θα τους υποχρεώσει να κάνουν το σωστό. Ο κύριος Αλάντ, ο οποίος είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Τατσαλήμ, λέει τον ΟΗΕ, στο Συμβούλιο Ασφαλείας τον Οκτώβριο του 2016, ότι το Ισραήλ δεν θα πάψει να είναι ο καταπιεστής εάν δεν υποχρεωθεί να αναλάβει τις ευθύνες για την ε, βιότητα της πολιτικής του. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Αυτοί οι Ισραηλινοί θέλουν τη βοήθειά μας και πρέπει να μας δουν στο πλευρό τους. Πολύ σύντομα, Υπάρχει οπτική γωνία των διεθνών πραγμάτων και των εσωτερικών. Το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να βασίζεται τις κατευθύνσεις αρχές που διέπουν και τη λειτουργία του ΙΕ. Γιατί αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σε σχέση με τους επικισμούς του Ισραήλ. Αυτά ω προ το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο. Τώρα στα εσωτερικά πράγματα και τη διαδικασία μια αναγνώριση. Υπάρχει ένα φάσμα κρατών και εταιριών ε, ευρωπαϊκών, αλλά και αλλού στον κόσμο. Υπάρχει μια σειρά από ζητήματα εγχώρια και εσωτερικά, τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά από το Συμβούλιο Ασφαλείας Χάρη του δηλαδή είναι η αδυναμία επιχειρηματιών να λάβουν δικαιώματα και να μπορέσουν να δράσουν ώστε να υπάρξει μια οικονομική ε, δραστηριότητα. Υπάρχουν σύμβουλοι από τουλάχιστον 17, 18 ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίοι έχουν εκφράσει προειδοποίησεις λέγοντας ότι οικονομικά, χρηματοπιστωτικά και νομικά ε, προβλήματα και απειλές ε, ελοχεύουν. Όλα αυτά που να μεταφραστούν σωστά σε μέτρα συμμόρφωσης για τις εταιρείες σε ιστορικό επίπεδο και για εφαρμαστικούς κανόνες για τα κράτη-μέλη και τις ε, αρχές του κάθε κράτους μέλους που θα πρέπει να διευθετεί τη δράση αυτών των επιχειρήσεων για να μην παίρνουν ας πούμε δικαιώματα και ωφέλη παρανόμως Κύριε Χάμαρπερκ ναι, πολύ σύντομα. Ε, σημειώνω ότι οι δύο εκπρόσωποι της Παλαιστίνης που είναι εδώ στην αρχή της διάσκεψης και οι δύο τελείωσαν τις ομιλίες τους λέγοντας ότι είστε ευπρόσδεκτοι να έρθετε να μα επισκεφτείτε στην Παλαιστίνη. Εδώ υπάρχει ένα διπλό μήνυμα. Διότι πρόσεξα ότι όλοι όσοι πάνε ως εκεί και έρχονται σε επαφή με ανθρώπου στην Ελλάδα τη Γάζα, αν μπορούν να μπουν ω εκεί και στη Δυτική Όχθη, έρχονται τελείω αλλαγμένοι πίσω, διότι βλέπουν την πραγματικότητα. Δεν μπορούν να τη δουν από τα μέσα μαζική ενημέρωση σπίτι του. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να μπορούμε να μιλάμε για την πραγματικότητα των καθημερινών ανθρώπων. Θα πρέπει να έχουμε τα κότσια να το κάνουμε αυτό όσο και αν μας καταθλίβει η κατάσταση της έννοιας της λύσης των δύο Εγώ είμαι εντελώ κατά της υπονόμευσης της προσέγγισης των δύο κρατών, είμαι εντελώ αντίθετος, διότι έχουμε μια διεθνή ε, συμφωνία ως προς την προσέγγιση των δύο κρατών. Εάν ε, κάνουμε μια προστοχώρηση προς αυτό, πού θα πάμε. Δηλαδή πάμε με το μέρος όσων δεν θέλουν λύση. Ε, ενώ λοιπόν ε, συμφωνώ με το συμπέρασμά σα, θα πρέπει να κοιτάξουμε την καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων στα καταχώμενα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ακριβώς την ώρα μας ολοκληρώθηκε αυτό το πάνελ. Θα ήθελα τώρα βάσει του προγράμματος να περάσουμε στον κύριο Ρίτσαρντ Φόκ και το βίντεο κλιπ του. Ευχαριστώ. Χαιρετίζω όλους όσους ε, παρίστανται σε αυτή τη διάσκεψη και θα ήθελα να σας εκφράσω τη θλίψη μου που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί σας για να συμμετάσχω ενεργά ε, και πλήρως στις σημερινές συζητήσεις. Είναι αναμφίβολο ότι τα πάνελ θα συνεισφέρουν ε, τα μάλλα και είμαι ευγνώμων από την άλλη μεριά που έχω την ευκαιρία παρόλα αυτά να πω δύο λόγια για το θέμα της σημερινής διάσκεψης και για το πώς εγώ ερμηνεύω το γεγονός ότι μετά από 50 χρόνια καταπιεστικής κατοχής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία ευκαιρία την οποία θα έπρεπε να είχε χρησιμοποιήσει πριν από χρόνια. Έχει παράλληλα αυτά μια ευκαιρία να ασκήσει μια κάποια πίεση στο Ισραήλ, ούτω ώστε να έχει μια πιο θετική προσέγγιση με σκοπό να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση και να δώσει δυνατότητα στους, στον Ισραηλινό λαό μετά από μια τόσο μακρά και δύσκολη εμπειρία να αποκτήσει τα θεμελιώδη δικαιώματά του. Πάνω απ' όλα το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση. Πιστεύω ότι αυτό ξεκινάει με την ελπίδα ότι θα υπάρξει κάποιο είδους μέλλον για τους Παλαιστίνιους που με βάση τα όσα προβλέπει και το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ήθος, ε, η διεθνής ηθική. Αυτό εξαρτάται από την αύξηση της εξωτερικής πίεσης ε, προς το Ισραήλ για να ξανασκεφτεί τα συμφέροντά του και να προωθήσει αξίες που υποτίθεται ότι δέχεται. Αυτή η διαδικασία Δούλεψε με πολύ αργό ρυθμό βέβαια στην Νότια Αφρική, αλλά τελικά οδήγησε τους ηγέτες της Νότιας Αφρικής να κάνουν αυτό που θεωρείται το Να ξεκινήσουν μια διαδικασία συμφιλίωσης με τον αφρικανικό πληθυσμό, που οδήγησε σε μια συνταγματική μεταρρύθμιση της χώρας, που στην αρχή είχε προβλήματα, αλλά τουλάχιστον οδήγησε στο τέλος του ρατσιστικού καθεστώτος του Απαρτχάιντ, που ήταν ενσωματωμένο και άρρηκτα δεμένο με την νότιο αφρικανική εμπειρία. Ε, τώρα βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε και να σκεφτούμε το θέμα της ε, κατοχής της Δυτικής Όχθης, της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και της Γάζας. Μετά από 50 χρόνια μετά από 50 χρόνια χρειάζεται κάποια φαντασία για να συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει στο λαό της περιοχής να ζει υπό μία ξένη στρατιωτική κατοχή για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ιδέα της Σύμβασης της Γενέβης, η τέταρτη Σύμβαση της Γενέβης για την εμπόλεμη κατοχή, ήταν ότι θα ήταν μια ε, διαδικασία προσωρινή, όπου οι δυνάμεις κατοχής θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους επί τη βάση της άσκησης μιας ελάχιστης παρέμφασης στα εσωτερικά του πληθυσμού, των αμάχων δηλαδή, ε, με έναν τρόπο που να μην αλλοιώνει τη φύση της κοινωνίας των πολιτών, που, μιας κοινωνίας που την έχουν υπό την κατοχή. Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η θεμελιώδη στόχη της τέταρτης ε, σύμβασης της Γενέβης και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου όλος ιδιαίτερος. Πρέπει να αποδοθεί κάποια δικαιοσύνη. Πρέπει να δούμε τις αντιφατικές πολιτικές και πρακτικές ε, που ζουν οι Παλαιστίνοι σε αυτές τις συνθήκες κατοχής. Καταρχάς, αυτή η κατοχή ε, έχει τραβήξει για μένα μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει ε, φως ε, στο τέλος του τούνελ. Όπως σας είπα, η Σύμβαση της Γενέβης προέβλεπε μία πολύ βραχυπρόθεσμη κατοχή, όπου οι συνθήκες για μια βιώσιμη ειρήνη θα είχαν υλοποιηθεί μέσα σε μια περίοδο που δεν θα ξεπερνούσε ας πούμε την πενταετία. Αυτή όμως η σημερινή κατοχή έχει ξεπεράσει το, την πεντηκονταετία και έχει μία σειρά από πολιτικές και πρακτικές που έχουν πλήξει την ποιότητα ζωής των Παλαιστινίων που ζουν υπ' αυτές τις συνθήκες στις τρεις ζώνες κατοχής. Η δυτική όχθη υπάρχει, στη δυτική όχθη μάλλον, υπάρχει καθημερινή παρέμβαση των Ισραηλινών με τα θέματα της ε, κινητικότητά τους. Ε, υπάρχει η ταπείνωση που ζουν οι Παλαιστίνοι με τα οδοφράγματα, με τα σημεία ελέγχου. Ε, ξαφνικές επιθέσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας των Ισραηλινών και ε, παρεμβαίνουν συστηματικά ε, στην προοπτική για ένα Παλαιστινιακό κράτος η Ισραηλινή ε, με το φαινόμενο των ε, επικισμών. με κατάφορη παραβίαση του άρθρου 49 παράγραφος 6 της 4ης Σύμβασης της Γενέβης που καταδικάστηκε από το ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας τον Δεκέμβριο του 2016. Το ψήφισμα αυτό ήταν σημαντικό γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, το Συμβούλιο Ασφαλείας ήταν σε θέση να πάρει μια απόφαση που, θα, που επέκρινε το Ισραήλ, όπου οι Ηνωμένε Πολιτείες αντί να ρίξουν, να, βάλουν βέτο όπως κάνουν συνήθως, ε, απήχαν. Θα μπορούσε να θεωρηθεί και πρέπει να θεωρηθεί ακόμα και τώρα ως ένα σημάδι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μια νέα προσέγγιση απαιτείται και μάλιστα έπρεπε να είχε προωθηθεί πολύ πιο πριν. Η κατοχή αυτή συνεχίζεται επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό δεν μπορεί να είναι πλέον ανοιχτή. Και το Ισραήλ δεν δείχνει, καμία, κανένα, δεν δείχνει κανένα σημάδι ότι είναι έτοιμο να αποσυρθεί. Έχει ενσωματώσει, έχει προσαρτήσει την Ιερουσαλήμ, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στο λεγόμενο στη λεγόμενη αιώνια πρωτεύουσα του Ισραήλ. Έχει κρατήσει το λαό της Γάζας σε ομοιρία με τις ανοιχτές αυτές φυλακές, όπου οι φυλακισμένοι περιοδικά υφίστανται μαζικές επιθέσεις. Και στην Δυτική Όχθη έχουμε εκτεταμένους επικισμούς ε, σε συνδυασμό με σημεία ελέγχου και με μία πολύ αβέβαιη καθημερινότητα, με μια πολύ αβέβαιη και ευάλωτη ζωή για τους Παλαιστίνους. Επίσης έχουμε τον κατακαιρματισμό της Δυτικής όφης μέσω των αρχικών ε, περιοχών Α, Β και Γ των συμφωνιών του Όσλο. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που μπορούμε να πούμε είναι ότι η κατοχή έχει παρατραβήξει για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ασκείται με έναν τρόπο που είναι ασυνεπής με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα πάρα αυτά. Όπως ε, είπε και ο ειδικό εισηγητής για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη στην πρόσφατη ε, συγκλονιστική έκθεσή του. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι η κατοχή από την ε, αρχή, το 1967, από την αρχή της, ποτέ δεν ε, δημιουργήθηκε ε, για να υλοποιήσει τους βασικούς στόχους της Σύμβασης της Γενέβης. Αντίθετα, έχει εξυπηρετήσει και έχει χρησιμεύει ως εργαλείο στους Ισραηλινούς για να υλοποιήσουν το όραμα για ένα, μεγαλύ... ένα Μίζων Ισραήλ, που το όραμα του σιωνιστικού κινήματος. Ε, στην, στο Ισραήλ ε, οι δυτικοί όχθη αναφέ, την, την, αναφέρουν ως Ιουδαία και Σαμάρια. Και εμείς, όπως σας είπα, το Ισραήλ έχει προσαρτήσει την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα εδάφη του. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι Η κατοχή θεωρείται από τη Σύμβαση της Γενέβης ως ένας προσωρινός τρόπος για να μεταβούμε από τον πόλεμο στην ειρήνη. Αντίθετα, εδώ στην προκειμένη περίπτωση, οι δυνάμεις κατοχής έχουν εδαφικές φιλοδοξίες. Και δεν κρύβουν το γεγονός ότι ο στόχος τους είναι να, να θεσπίσουν ένα μόνιμο έλεγχο κάποιου τύπου ο, επάνω σε όλα ή τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι, αν όχι σε όλο, της Δυτικής Όχθης. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουν να υλοποιήσουν πλήρως όλες τις ιονιστικές φιλοδοξίες, ούτως ώστε να υλοποιηθεί η βιβλική άποψη για το Ισραήλ. Αυτή η έννοια της κατοχής ήταν ένα προπέτασμα πίσω από το οποίο κρύβει το Ισραήλ τις πραγματικές προθέσεις του. Σε αυτή τη φάση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει το δικαίωμα να αγνοεί αυτές τις πραγματικότητες και θα πρέπει να λάβει βήματα που θα δείχνουν ότι αναγνωρίζει την πραγματικότητα και θα πρέπει να ασκήσει επαρκή πίεση, ούτω ώστε να βοηθήσει το Ισραήλ και έμεσα τις Ηνωμένε Πολιτείες και την κυβέρνησή τους να προβούν στις απαραίτητες προσαρμογές, ούτω ώστε να ε, φτάσουμε σε μία δίκαιη ειρήνη για τους δύο λαούς. Κάτι που σημαίνει το να τεθεί τέρμα στις προσαρτήσεις από πλευράς Ισραήλ, καθώς και να διαλυθούν, να διαλυθεί αυτή η δομή του apartheid, μέσα στην οποία ο λαός του, της Παλαιστίνης είναι θύμα λόγω της φυλής του. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή είναι μια νέα μορφή apartheid. Θα σας ε, αφήσω τώρα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία σε αυτές τις συζητήσεις και ελπίζω ότι όλες αυτές οι συζητήσεις θα αυξήσουν την παγκόσμια αλληλεγγύη για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και θα βοηθήσουν στο να επέλθει τελικά η ειρήνη μεταξύ των δύο αυτών λαών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Φακ για την ε, σύνοψη αυτής της συζήτησης. Εδώ δεν θα έχουμε ερωτήσεις, σχόλια και παρατηρήσεις. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους εξαιρετικούς μας συμμετέχοντες στο πάνελ. Ήταν φανταστική παρασίαση αυτού του προβλήματος που δεν έχει τέλος. Θα ήθελα εδώ να προσκαλέσω τους επόμενους συμμετέχοντες στο πάνελ με την Προεδρία της συναδέλφου και μέλους ε, της Αντιπροσωπής για την Παλαιστινή της κυρίας Άουκεν Καλησπέρα σας. Θα συνεχίσουμε να περάσουμε στο δεύτερο πάνελ τώρα. Ο κύριος Ότε. Θα περάσουμε στα πολιτικά θέματα τώρα. Αν έχετε τίποτα καινούργιες ιδέες για να το πώς θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ως τώρα παθητική στάση και θα ήθελα να σας κινητοποιήσω για να μου πείτε τα μηνύματά σας που μπορεί να είναι και λίγο δυσάρεστα ίσως δεν θα επαναλάβω τις συστάσεις, τα βλέπετε με λεπτομέρειες όλους τους τίτλους στο χαρτάκι σας που έχει το πρόγραμμα. Παρακαλώ, λόγο σε εσάς. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ζητήσω συγγνώμη για την φωνή μου. Είχα ένα άσχημο κρυολόγημα και παρόλα αυτά ελπίζω συνεχίσετε να με καταλαβαίνετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είχα την τύχη να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, καλή ή κακή, για πολλά χρόνια. Μιλάμε για 50 χρόνια κατοχής. Αυτά τα 50 χρόνια είναι το αποτέλεσμα μιας ανεπίλητης ε, διένεξης που αρχίζει από πολύ παλιότερα βέβαια. έχει να κάνει και με την απόφαση του ΙΕ για τη Βρετανική εντολή προστασία της Παλαιστίνης και το ψήφισμα 181 του 1947 το οποίο ε, προβλέπει τη δημιουργία αραβικού και εβραϊκού κράτους. Αυτό απερίφθη από τους Άραβες και αυτές είναι οι συνθήκες που οδήγησαν στον πόλεμο. Τον πόλεμο μεταξύ κρατών Εντό κρατών με τρομοκρατικές, σεκταριστικές και εξτρεμιστικές δράσεις ε, πολλές φορές ε, με άλλους να εκπροσωπούν τα συμφέροντα των και των δε. Τώρα βλέπουμε πως έχει δημιουργηθεί, ε, τι κατάσταση έχει δημιουργηθεί στη Λωρίδα Τριγάζα, στη δικαιώθηκε και εντός και εκτός Ιερουσαλήμ βλέπουμε να υπάρχει μια τελείως διαφορετική αφήγηση ε, από πλευράς Αράβων και Εβραίων. Ε, με τελική φάση της ε, σύραξης ενδεχομένως να παίρνει μέρος και το Ιράν για να επιλύσει το θέμα, η Τουρκία. Ε, από το 1967 ε, φαίνεται να είναι η στιγμή για τη δημιουργία μιας νέας τάξης στη Μέση η στιγμή αυτή. Όμως αυτό ίσως όδευε από πολύ καιρό προς εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεχτεί κατά κάποιο τρόπο ότι η ανεπίλητη διαφορά είναι μεταξύ Ισραηλινών και Αράβων, όχι Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Ούτως ή άλλως, διαρκώς οι Άραβες κατηγορούν για την απουσία προόδου προς τη λύση των δύο ε, κρατών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Άραβων και Ισραηλινών δεν ήταν άμεσες και δεν έχουν πετύχει. το να υπάρξει νόμιμη διαδικασία και να δεσμευτούν και τα δύο μέρη, ο δικό χάρτη και η σωστή προσέγγιση θα ήταν συνθήκε για να μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να δημιουργήσουν το δικό του κράτο με δικά του μέσα και θεσμού. Ο Πρωθυπουργό Φαγιάντ ζήτησε την βοήθεια και των Ευρωπαίων, ενώ οι Ισραηλινοί σιωπηρά δέχτηκαν την παροχή βοήθεια, κυρίω στον τομέα τη οικονομία και των υποδομών. Όμως υπάρχει καχυποψία και από τις δύο πλευρές, τις δύο μπλεκόμενες πλευρές και δεν έχει βρεθεί ακόμη λύση. Ο βασικός διαμεσολαβητής ε, τελικά προσπαθεί να εξομαλύνει απλώς αυτές τις ασυμμετρικές σχέσεις, αλλά αυτό μειώνει πολύ το περιθώριο μόχλευσης. Όπως δείχνουν και τα πρωτοσέλιδα, τα τελευταία 50 χρόνια η κατοχή αυτή ε, οδηγεί στο εξή και μόνο συμπέρασμα. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Αυτό είπε ο υπατός και αυτό αποσχέθηκε να κάνει μετά την ε, συνάντηση με τους υπουργούς εξωτερικών στο Τάλιν όπου έγινε λόγος για την απουσία προόδου. Εκεί η είπατε πρόσωπος είπε ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε την ε, πίεση για να επιτύχουμε πολιτικούς στόχους. Η ευρωπαϊκή πολιτική είναι πολύ πολύπλευρη και έδρη σε σχέση με την ε, διαφορά αυτή. Έχει απεικονιστεί από δηλώσεις στη Βενετία, το Βερολίνο, ε, με διπλωματικές οδούς προς τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές, προς διεθνείς πρωταγωνιστές και φορείς, ε, ε, με πρακτικό περιεχόμενο, με διεθνές χαρτοφυλάκιο το μεγαλύτερο για την υποστήριξη των Παλαιστινίων, με ανθρωπιστικές προεκτάσεις, με την ε, προσπάθεια στήριξης της οικοδόμησης θεσμών από τους Παλαιστινίους, με την αναγνώριση ότι οι Παλαιστίνοι είναι έτοιμοι να έχουν ένα κάτω που θα λειτουργήσει όσο το δυνατόν συντομότερα, μόλις βρεθεί μια πολιτική συμφωνία και υπογραφή αυτή. Από την άλλη, ανοίγει η προοπτική για το Ισραήλ να έχει μια ισχυρή εταιρική σχέση, σχέσει ε, συμφωνίε και συνεργασία σε τομεί όπω το εμπόριο, η τεχνολογία, οι επιστήμε, ε, η ασφάλεια, για την ε, τάση ειρήνευσης ε, στο, στις περιοχές που μοιράζονται με τους Παλαιστινίου και για να υπάρξει με προπόθεσμα η αναζήτηση της ειρήνης με τον αραβικό κόσμο. Δεν μπορούν να αλλάξουν τελείως οι αρχές που διέπουν αυτή την ε, κατοχή και τρόποι δράση, αλλά πρέπει να αλλάξουν οι τρόποι με τους οποίους όλα αυτά εφαρμόζονται. Θα πρέπει το στρατηγικό περιβάλλον στην περιοχή να το δούμε με άλλο τρόπο και να αντλήσουμε διδάγματα από τις ε, δράσεις του παρελθόντος. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε την αίσθηση ότι αυτή η τάση σύγκληση στατικών συμφερόντων μεταξύ Ισραηλινών και γειτόνων του μπορούν να ε, ε, χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν κοινέ διεθνεί απειλέ, όπω η απειλή της του τζιχάντ, η διεθνή τρομοκρατία. Θα πρέπει επίση να υπάρξει επιχειρηματική πρόοδο. Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δοθεί τέρμα στην κατοχή και να αναγνωριστεί να αναγνωριστούν τα εθνικά δικαιώματα των Παλαιστινίων ε, όπω εκφράζονται από το Διεθνέ Δίκαιο. Θα μπορούσε να υπάρχει νομιμοποίηση στη συνεργασία του Ισραήλ με την κοινή γνώμη των αραβικών κρατών που είναι πολύ ευαίσθητε σε σχέση με το με το δράμα που ζουν οι Παλαιστίνοι. Θα πρέπει να υπάρξει πρακτική εφαρμογή των όσων προβλέπουν τα ψηφίσματα τη Γενική Συνέλευση και του Συμβούλου Ασφαλεία του ΟΗΕ. Και μάλιστα πρακτική εφαρμογή τη ε, πρωτοβουλία για την ειρήνη των ε, Αράβων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει νέα όθηση σε αυτήν την πολυμερή προσέγγιση και οδό εξέβριση λύση μα στη διαδικασία τη Βακελόνη, προσπαθώντα να επιβάλλει ένα νέο καθεστώ για την ειρήνη. Ο ευρωπαϊκός ρόλος ε, στην ε, συμφωνία με το Ιράν, ο πολιτικός διάλογος με την Τεχεράνη θα μπορούσε να δώσει ένα διευκολυντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξέβεση λύσης γενικότερα, ώστε να αντιμετωπιστεί και το πραγματικό πρόβλημα των Παλαιστινίων. Επίσης, η ειρηνευτική διαδικασία που ανακοινώθηκε τον πρόεδρο Τραμπ θεωρούμε ότι μπορεί να αρχίσει να επιχειρείται από τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να συμμετάσχουν πλήρως και να πείσουν τους Ηνωμένε Πολιτείε για τις υποχρεώσεις και τις δυνατότητες που μπορεί να αναπτύξει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον η ευρωπαϊκή στήριξη θα μπορούσε να τονώσει την νομιμοποίηση της αμερικανικής προσπάθειας. Τρίτον, αρνητικές τάσεις που έχουν επιπτώσεις και στις κοινωνίες και τις κοινωνίες των πολιτών. Δεν μπορεί η σημερινή κυβέρνηση που δεν υποστηρίζει τη λύση των δύο κρατών να παραμείνει ε, έχει. Δεν μπορεί να προωθούνται συμφέροντα που είναι απαράδεκτα για την άλλη πλευρά και να ε, διακυβεύεται η ασφάλεια και η ειρήνη οι επικισμοί στα κατεχόμενα πρέπει να πάυσουν εφόσον καθιστούν άκυρη την ε, εξέβρεση λύσης δύο κρατών. Θα πρέπει η δημοκρατία ε, να προστατευτεί και να μην υπάρχουν εξτρεμιστικές σεκταριστικές ε, και ε, Θα πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση και στις Βρυξέλλες με τις επισκέψεις πολιτικών ηθινόντων και να δούμε ποιες είναι οι καλύτερες δυνατές συνθήκες που μπορεί να βρεθούν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργό είπε ότι έχει χάσει... Ο Παλαιστίνιος μάλλον ε, Πρωθυπουργός είπε ότι έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της νομιμοποίησής του εναντί της κοινής γνώμης και κυρίως των νέων με την πρόσφατα γεγονότα. Από το 2016 εντοπίζεται ότι 14%, 48% θα ήθελε να διαλυθεί η αρχή, η ανεξάρτητη αρχή των Παλαιστινίων. Ε, στην Παλαιστίνη η κατάσταση των νέων χειροτερεύει. Ταυτόχρονα η κοινωνία των ε, Παλαιστινίων ρωτήστε δυναμικά, δείχνοντα τι δυνατότητε έχει η κοινωνία των πολιτών. Είναι πολύ ε, καλά διασυνδεδεμένη η Παλαιστίνη και δείχνει αυτό πόσο ε, οι αραβικές κοινωνίες είναι ευαισθητοποιημένε για τα θέματα των δικαιωμάτων. οι Παλαιστίνοι θα μπορούσαν να αναπτύξουν και πολιτική δράση εντό του ε, Ισραηλινού συστήματο. Αυτά θα εξυπηρετούσαν την κοινωνία των πολιτών και τι επιχειρήσει. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στου ηγέτε τη Φατάχ και τη Χαμά για να λάβουν υπόψη τι ανάγκε διεθνού προσπάθεια για να επιτευχθεί πρόοδο, ακόμη και με τη τη Αιγύπτου. Θα πρέπει να πάψει η κατοχή και να υπάρξει εθνική αυτοδιάθεση και ανεξαρτησία. Επίση, πρέπει να ξαναδούμε πώ ε, εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με αυτή τη διαφορά για να προσαρμοστούμε και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο πλαίσιο των ε, τοπικών και διεθνών εξελίξεων. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή μόχλευση να αξιοποιηθεί και να μπορέσει να λάβει σε η ευρωπαϊκή δράση. πρέπει να υπάρξουν παράλληλοι δρόμοι και όχι διαδοχικά στάδια προς το παρελθόν, αλλά πρέπει να δώσουμε έμφαση στα, στην περιφερειακή και πολυμερή διάσταση και θα πρέπει όσα συμφωνούνται να εφαρμόζονται αμέσω. Διότι αλλιώ ε, ισχύει το δίκαιο του ισχυροτέρου. Και θα πρέπει προσπάθειες προκολούθησης να αναλυθούν από τη διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Οτέ. Και τώρα... Θα ήθελα να μιλήσουμε πιο διεξοδικά για αυτή τη στρατηγική. Και ακριβώς γι' αυτό θα δώσω το λόγο στον Μπιχάρα Κάντερ. Θα ήθελα να ακούσω τη δική του συνεισφορά. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, Δεν ήρθα σε αυτή τη διάσκεψη χωρίς τίποτα στα χέρια μου. Ετοίμασα μια ειδική έκθεση 35 σελίδων με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το θέμα της Παλαιστίνης 1957 μέχρι 2017». Ελπίζω ότι θα διανεμηθεί αυτή η έκθεση. Είμαι σίγουρη ότι αν δεν έχει μοιραστεί τώρα, θα μοιραστεί μαζί με τις υπόλοιπες ε, εκθέσεις των συναδέλφων μου. Δεν θέλω να κάνω αναδρομή στην ιστορία. Έχω, έχω γράψει ένα βιβλίο 700 σελίδων ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Παλαιστίνη από την εποχή της Σταυροφορίας μέχρι σήμερα. Ε, αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η Σταυροφόροι, η αποστολή και η εκστρατεία του, Ναπολε... του Ναπολέοντα συγγνώμη, Η συμφωνία του 16, η δήλωση του Μπαλφούρ του 17, ε, η οργάνωση των Βρετανών από το, των Βρετανών από το 22 και μετά και η δημιουργία του Ισραήλ μετά την ε, διέρεση, την οποία υπερψήφισε η Ευρώπη το 1947. Η Ευρώπη είναι υποχρεωμένη να αναλάβει τις ιστορικές ευθύνες απέναντι στην Παλαιστίνη και στον Παλαιστινιακό λαό. Από το 1948 και μετά, οι Ευρωπαίοι γενικά ε, συντάσσονται στο πλευρό των ε, Ισραηλινών. Έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν την ύπαρξή τους. Για να τους ε, απομονώσουν και να τους προστατεύσουν από τους Άραβες γείτονες και να τους ε, υποστηρίξουν οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά. Η σημαντική, η στρατηγική σημασία του Ισραήλ τονώθηκε. Ε, δεν είναι μόνο ένας ασφαλής ουρανός, αλλά και ως ε, προμαχώνας ε, που προστατεύει τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα απέναντι στους Άραβες. Αυτό σήμαινε παράλληλα κατακαιρματισμό των εδαφών μας και εκτοπισμό των λαών μας. Αυτό θεωρήθηκε από τους Ευρωπαίους ως παράπλευρη απώλεια. Και το παλαιστινιακό θέμα αντιμετωπίστηκε ως θέμα ανθρωπιστικό και ως θέμα προσφύγων. Από το 1967 η ευρωπαϊκή θέση αλλάζει όμως. Το παλαιστινιακό θέμα αναβαθμίζεται. 1973. Οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν τις, ε, τα νόμιμα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Το 1947 το 1974, συγγνώμη, ε, η ανάγκη για την πατρίδα των Παλαιστινίων. Στη δήλωση της ε, Βενετίας το 1980 ε, ζητείται μια ειρηνική λύση της σύγκρουσης με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις του PLO. Αργότερα στη Μαδρίτη αναγνωρίζουν ότι το PLO θα πρέπει να συμμετέχει 100% στις διαπραγματεύσεις. Το 1999, όταν ο Αραφάτ ήθελε μονομερός να δηλώσει το Παλαιστινιακό κράτος όπως προβλεπόταν στι συμφωνίες του Όσλο, η Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε πίεσαν τον Αραφάτ να μην κάνει αυτή τη μονομερή ε, ανακήρυξη και στην δήλωση του 1999 ε, του υποσχέθηκαν ότι θα αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος ε, εν ευθέτω χρόνο. Ακόμα περιμένουμε. Και όμως η Ευρώπη θεωρεί ότι το Ισραήλ είναι πρωτεύουσα και του Συγγνώμη ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι η Ιερουσαλήμ είναι πρωτεύουσα και του Ισραήλ και της Παλαιστίνης. Αυτή η πολιτική του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θεωρείται ως μια διπλωματία μεγάφωνο, ε, μια προκατηλημένη θέση. Η δική μου, έτσι λένε οι άνθρωποι στην περιοχή, εγώ θεωρώ ότι παρά τις ασυνέπειές της, η Ευρώπη, δηλώνοντας την, ότι είναι νόμιμη η προσάρτηση, κατοχή. Συγγνώμη, ότι είναι παράνομη, στην πραγματικότητα συνεισέφερε ε, στο να αναδειχθεί ως νόμιμο το αίτημα των Παλαιστινίων για ένα κράτος. Παράλληλα, επειδή στην πραγματικότητα παίζει το δεύτερο βιολί στα όσα κάνουν οι ΗΠΑ... και επειδή είναι το παραπέδι στις, ε, στις διαδικασίε, διαδικασίες και απλώς ε, βοηθά οικονομικά τους Παλαιστίνιους ε, εν μόνιμης και βιώσιμης λύσης, αφήνοντας τις Ηνωμένε πολιτείες να κάνουν παιχνίδι με τραγικές συνέπειες, καταστρέφοντας τα κατεχόμενα εδάφη, όπως μας είπε ο, Ρίτσαρντ και με προσαρτήσεις, όπως μας είπε ο Τόμας επίσης, η Ευρώπη έμεσα διατήρησε την, και βοήθησε στο να συνεχιστεί η κατοχή της Παλαιστίνης. Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην πραγματικότητα και στη ρητορία. Αυτή η αποτυχία δεν είναι ε, το αποτέλεσμα της, του ευρωπαϊκού αφηγήματο, αλλά των διαφορετικών πολιτικών και μνημών και απόψεων που έχουν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ε, λόγω των θεσμικών της περιορισμών. Πολλά από τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πήγαν ε, και αποδυναμώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι και η ώρα να αλλάξει πορεία η Ευρωπαϊκή Ένωση, να αλλάξει μέσα, να αλλάξει μέθοδο και να καταλάβει πλήρως ποιο είναι το εύρος του Παλαιστινιακού προβλήματος. δεδομένου του μόνιμου προβλήματος των Παλαιστινίων, τον, τον άκμπα το λεγόμενο, το αδιέξοδο, ε, από το 47 μέχρι σήμερα, δεδομένης της, ε, του γεγονότος ότι η σύγκρουση αυτή έχει επιπτώσεις σε όλη την περιοχή, λόγω του γεγονότος ότι Υπάρχει μια εξωτερικοποίηση της σύγκρουσης αυτής λόγω της, ε, του, του μόνιμου δηλητηρίου που, και αγκαθιού που αποτελεί το Παλαιστινιακό στην περιοχή αυτή, το να επιληθεί η σύγκρουση αυτή, δεν είναι απλώς προς το συμφέρον των Παλαιστινίων μόνον, αλλά και είναι και προς το συμφέρον και των Ισραηλινών και των Δυτικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι χαλαρές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, η, η άνοχή της απέναντι στους Ισραηλινούς θέτουν να την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι έτσι, δεν λειτουργεί έτσι ένας αξιόπιστος γεωπολιτικός παίχτης στην ε, άμεση γειτονία του. Η οικονομική βοήθεια είναι σίγουρα επίγουσα και απαραίτητη και οι Παλαιστίνοι είναι ευγνώμονε για τη βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε για να υποσκάψετε την αντίσταση των Παλαιστινίων ή να δικαιολογήσετε την κατοχή. Η Ευρώπη θα πρέπει να υποστηρίξει αυτή την τρίτη η ειρηνική Ιντιφάτα, όπως είπε και ο Τόμας Φρίντμαν ε, από το New York Times πριν από λίγους μήνες, που είναι μια εκστρατεία που δεν θέλει να απονομιμοποιήσει το Ισραήλ, αλλά την κατοχή του και τις πολιτικές του. Επομένως, η η στυλίτευση από κάποιες ε, ευρωπαϊκές χώρες της Ιντιφάντας αυτής στην πραγματικότητα είναι επιζήμια για τον Παλαιστινιακό λαό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει του Ισραηλινούς να καταλάβουν ότι τελείωσε η εποχή της ατιμορρησίας ε, και δεν υπάρχει καθόλου και πουθενά κατοχή χωρίς κόστος. Το να ε, το να βάζουμε ετικέτες, Ισραηλινά προϊόντα από, τα, από τους επικισμούς, δεν αρκεί αυτό. Όταν ε, η, η Ρωσία άρχισε να εξάγει προϊόντα από την Κρυμαία, η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι θα πρέπει να σταματήσει το εμπόριο με προϊόντα από την Κρυμαία. Το ίδιο θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια προϊόντα που δεν θα πρέπει να μπαίνουν σε ευρωπαϊκές αγορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πει ότι η πολιτική των επικισμών του Ισραήλ με την, η προσάρτηση της Ιερουσαλήμ, ο κατακαιρματισμός των εδαφών μας, καθιστούν την ε, λύση των δύο κρατών γεωγραφικά αδύνατη. Πώς μπορεί η Ευρώπη να μιλήσει για μια βιο, ένα βιώσιμο, συνεχές, ανεξάρτητο κράτος υπ' αυτές τις συνθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη σύστασή της, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τη σύστασή του μάλλον, ε, ζήτησε ε, να, υπάρξουν αυτές, να υπάρξει αυτή η λύση των δύο κρατών, αλλά έχουν αγνοηθεί αυτές οι συστάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να ζητήσει την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους με ή χωρίς διαπραγματεύσεις. Όπως προτείνει ο πρώτος ανεσταλμένος ο κύριος Μορετίνο στην ε, Μέση Ανατολή. Και την περασμένη εβδομάδα ακόμα υπόθηκε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αναγνωρίσει πάρα αυτά το κράτος της Παλαιστίνης, χωρίς διαπραγματεύσεις. Και ο, ο, Χουριών το 1948, ούτως ή άλλως, ο Μπεν Χουριών, ε, δια, ανακήρυξε το κράτος του Ισραήλ ε, μόνο, μονομερός. η επίκριση των ε, πολιτικών του Ισραήλ δεν είναι αντισημιτισμός. Το να επικρίνεται ε, τις ε, Ισραηλινές πολιτικές και να με αντισημιτισμό, στην πραγματικότητα φημώνεται την, την νόμιμη κριτική. Και αυτό υποσκάπτει την ε, ελευθερία έκφρασης. Τέλος. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να πάψουν να θεωρούν το Ισραήλ μία εξαίρεση. Δεν υπάρχει πουθενά ε, στο εθνικό δίκαιο ή στο δίκαιο ε, κάποια διάταξη που λέει ότι το Ισραήλ είναι τόσο εξαιρετικό πια που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε τελείως διαφορετικά από όλα τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank you. I wish... Πολύ σας ευχαριστώ. Μακάρι να εκπροσωπούσε εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν ευκολότερο να πω ναι, θα γίνει. Πάντω, από ό,τι βλέπω εδώ, εκπροσωπούνται πολλέ από τι πολιτικέ πτέρυγε του Κοινοβουλίου με τα μέλη που είναι παρόντα. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο λοιπόν μπορούμε. Τελευταίο θα δώσω το λόγο στον κύριο Χιου Λόβατ. Ανυπομονούσαμε, γιατί θα μα πείτε γίνεται για τα θέματα του διαχωρισμού και της διαφοροποίησης. Ξέρω ότι η δουλειά σας υπήρξε πολύ χρήσιμη σε σχέση με τα θέματα αυτά. Κάποιες από τις συστάσεις σας ήδη υλοποιούνται. Και με τις καλές σας συμβουλές πιστεύω ότι θα μας διαφωτίσετε. Ευχαριστώ και θα συνεχίσω από εκεί που έπαυσε ο Μάρκ Ότ. Όπως λέει, είπατε εκπρόσωπος Φεντερίκα Μογερίνη για την ε, συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και εμεί να οδεύσει. Ήταν ένα βήμα που χρειαζόταν εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα διακαώς. Και πέρα από την ε, στενή τεχνική επικέντρωση τη προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη οικονομική βοήθεια προ του Παλαιστινίου, θα πρέπει να υπάρξει μια σφαιρικότερη προσέγγιση των όσο συμβαίνουν εκεί. Να υπάρξει δηλαδή μια γενικότερη ανανέωση στην ευρωπαϊκή πολιτική, γιατί χρειάζεται μια σωστή διάγνωση τη όλη κατάσταση και χάραξη νέα πολιτική. Τη διάγνωση την ακούσατε σήμερα. Δυστυχώ, μπορεί να πει κανεί ότι στην Ουάσιγκτον και σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες τα συμπεράσματά τους δεν είναι τα με τα δικά μα σήμερα. Δηλαδή και 25 χρόνια γυρνάνε γύρω από την ουρά τους. Και κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν. Θα έλεγα λοιπόν, για να συνοψίσω λίγο τα όσα υπόθηκαν εδώ σε σχέση με την ακρίβεια της διάγνωσης που θα πρέπει να ε, ε, γίνει για την ευρωπαϊκή πολιτική, είναι κάτι που θα ευνηδιάζει του περισσότερου, αλλά το γνωρίζουν ότι η ενεργειακή διαδικασία του Όσλο για τη Μέση Ανατολή δεν έχει δώσει αποτελέσματα. Και εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε κατά πόσο προσπαθούμε να βάλουμε σε διαφορετική θέση τα έπιπλα μέσα στον τιτανικό που βυθίζεται. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φαίνεται να υποστηρίζει την λύση των δύο κρατών, κάτι που όλοι ε, θελήσαμε. Δεν δίνει μια αποφασιστική όθηση προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι εάν οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συνεχίσουν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να του αντικαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Κάτι που είχε κάνει για πολλέ δεκαετίε, του παραχωρήσει την θέση τη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Επίση, είναι σημαντικό η αδυναμία των Παλαιστινίων να σημειωθεί. Είναι και αυτό ένα μέρος της ασύμετρης αυτής ε, διαφοράς μεταξύ κατεχόντων και κατεχομένων. Είδαμε την εδαφή, τον εδαφικό και πολιτικό κατακαιρματισμό της Παλαιστίνης, αλλά επίσης, νομίζω ότι μπορεί να το πει κανείς εδώ, ότι κάπως ε, δημιουργείται ένας δημοκρατικός αυτό στην Παλαιστίνη, αλλά με συρρήκνωση τη συμμετοχή των πολιτών ε, στην δυτική τουλάχιστον όχθη. Όχι μόνο λόγω τη δράση των Ισραηλινών, αλλά και τη Παλαιστινική αρχή. Ο Κίτσαν Άντρο, ο οποίο ε, έχει έρθει και έχει μιλήσει εδώ, έχει φυλακιστεί. Η υπόθεσή του είναι μοναδική. Αυτό έχει αρνητικέ επιπτώσει ε, στην δραστηριοποίηση των Παλαιστινίων. Μειώνεται η αποτελεσματικότητα της δράσης τους, της στρατηγικής που θα μπορούσαν να χαράξουν για να αντιμετωπίσουν την κατοχή. Και το κατά πόσον εμείς μπορούμε να απευθύνουμε τις πολιτικές μας λύσεις προς αυτούς χωρίς να το λάβουμε υπόψη ως στοιχείο. Πρέπει δηλαδή να τα σκεφτούμε λίγο κι εμείς. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε τη δυνατά σημεία του Ισραήλ. Τα γνωρίζουμε βέβαια, αλλά έχει κύρος στην όλη περιοχή του Ισραήλ και αυτό διαρκώς αυξάνεται με ταχύς ρυθμούς. Είναι μια διαδικασία εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα κράτη του κόλπου, κάτι που πραγματικά έχει επιταχυνθεί και διαρκώς έρχεται επιτάπητος. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ίσως να υπονομεύσει τη διαδικασία την ειρηνευτική των Αράβων. Ο αλλά Δεν μα έδωσε του πώ αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Το Ισραήλ πάντως κοιτάζει με προσοχή τι συμβαίνει στον αραβικό κόσμο και το ζήτημα είναι τι δίνει ω αντάλλαγμα για την πρόοδο αυτή που επιτελείται. Η απάντηση ω τώρα είναι πολύ λίγα. Και μετά έχει σημασία για το διεθνέ προσκήνιο. Είδαμε την ανάδυση των ε, δεξιών ε, ακραίων κομμάτων των λαϊκιστικών κομμάτων που έχουν διαφορετικές ε, τοποθετήσεις σε σχέση με την διαφορά αυτή τη διάσταση από ό,τι ως τώρα έχει θετήσει η διεθνής κοινότητα ω τάση. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το διεθνές δίκαιο μπορεί να εφαρμοστεί διαφορετικά. Οι διεθνεί δεσμεύσει για την εξέβρεση λύση στην διαφορά μπορεί διαρκώ να διαβρώνονται λοιπόν. Το Ισραήλ στην Ευρώπη έβρισκε διαρκώς ομοειδεάτε του και σε αυτούς βασιζόταν. Έτσι προχώρησαν τα σχέδιά του και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, του έδινε το περιθώριο. και βεβαίω παρέμενε στην ατιμορρησία τη μη συμμόρφωση με τι διεθνεί υποχρεώσει και τι διεθνεί συστάσει. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε. Δεδομένη αυτή τη διάγνωση και εφόσον είναι σωστή, και σε σχέση με όσο είπε και ο καθηγητή Λίνκ και η δόκτωρ Αζάροβα και οι υπόλοιποι, Νομίζω ότι κατά πρώτον υπάρχει ανάγκη να αλλάξουμε το αφήγημα, τα όσα λέμε σε σχέση με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να μιλάμε απλώ για κατοχή. Πρέπει να μιλάμε για κατοχή που παίρνει τα χαρακτηριστικά τη προσάρτηση, το λιγότερο που μπορεί να πει κανεί. Υπάρχει ανάγκη ακριβού περιγραφή τη πραγματικότητα ω έχει, τη νομική πραγματικότητα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παράνομη διαρκού κατοχής. Δεν μπορούμε να, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε ε, την αρχική, το αρχικό κίνητο της δράσης των Ισραηλινών και να θεωρούμε ότι κάπως μαγικά θα περάσει αυτό διάθεση στα χέρια των Παλαιστινίων από τη μια στιγμή στην άλλη. Εδώ μιλάμε για πραγματική παραβίαση του δικαίου ε, για τον πόλεμο, bellum, και της χρήσης βίας. Εδώ οι υποχρεώσει των τρίτων κρατών είναι να απαιτήσουν να δοθεί τέρμα σε αυτή την κατοχή. Το Ισραήλ μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι πλέον ένας ένομο ε, κατέχων τη ε, Παλαιστίνη και των αδαφών τη. Πρέπει λοιπόν να αναλυθούν ευθύνε και από τα τρίτα κράτη και να παρέμβουν. Τι μπορούν να κάνουν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε εδώ ότι υπάρχει ένα όριο ε, σε σχέση με το ότι έχουν τη διάθεση να σκεφτούν ως πιθανές δράσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέλη της. Το μποϊκοτάζ κατά το Ισραήλ δεν είναι μεταξύ των επιλογών, ούτε η απαγόρευση εισαγωγή προϊόντων από τα κατεχόμενα. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να αποφανθούμε τώρα αν θα αλλάξει κάποτε ή όχι, αλλά ας κοιτάξουμε ποιε είναι εναλλακτικέ για να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε λίγο τον υπολογισμό των διασταυρούμενων ωφελών που θα μπορούσε να αντλήσει κανείς. Και να δούμε γιατί θα γινόταν αν εξακολουθήσει η σημερινή κατάσταση. Η εναλλακτική στη λύση των δύο δεν θα είναι η λύση του ενός κράτους, τουλάχιστον όχι σύντομα. Εάν όμως ε, ε, σβηστεί η λύση των δύο κρατών, θα είναι περισσότερο από τα ίδια που έχουμε ζήσει ως σήμερα. Περισσότερη προσάρτηση, περισσότερες ε, διαθέσεις καταστολής και καταπίεσης των Παλαιστινίων και το καθεξής. Με αυτά κατά νου λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ποιο θα είναι το όφελος εφόσον δέναμε τα χέρια μας για των Παλαιστινίων και οι Παλαιστίνοι δεν μπορούν να ζητήσουν ε, να υπάρξει διεθνής λογοδοσία, να μην πάνε στο διεθνές δικαστήριο, να μην ζητήσουν να καταγραφή των επιχειρήσεων σε κατάλογο, μαύρο κατάλογο όσων εμπλέκονται στους επικισμούς. Έπειτα, ενώ οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν φαίνεται ότι έχουν διάθεση να προσπιστούν τη λύση των δύο κρατών, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ότι μπορεί να το κάνει και μάλιστα και αποτελεσματικά. Αναφερθήκατε στα μέτρα διαφοροποίηση που απαιτούνται και το διεθνέ δίκαιο τα έχουν δοκιμαστεί. Ακόμη όμως εφαρμόζονται πολύ λίγο και περιορισμένα. Πολύ αργά μάλιστα. Το θέμα δεν είναι απλώς να παραμείνουν τα όρια του 67, τα πράσινα όρια του, η πράσινη γραμμή του 67 για τα όρια του Παλαιστινικού κράτους, αλλά και οι Ισραηλινοί να μαζέψουν τους επικισμούς τους και εντός και εκτός των ορίων τους. Και βεβαίως ε, να υπάρξει πίεση για τα όσα λένε εσωτερικός Ισραηλινοί για τις αυξανόμενες ε, δυσκολίες του προγράμματος επικισμών ε, για το πόσα ε, προβλήματα αντιμετωπίζουν και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε και την εμπάθηση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο πράγματα είναι ίσως σημαντικά, ίσως και λίγο περισσότερα. Ένα από τα μεγάλα σημαντικά βήματα στην προσπάθεια διαφοροποίησης ξεκίνησε το 2005, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ συμφώνησαν να αποκλείσουν τα προϊόντα των περιοχών του επικισμού από, την από τα τους προτιμησιακούς δασμούς. Από τότε που άλλαξε αυτή η πολιτική, φαίνεται ότι πάλι παίρνουν του προτιμησιακού δασμού τα ελληνικά προϊόντα του επικισμού. Να ένα πρόβλημα. Εδώ το Ευρωκοινοβούλιο μπορούσε να έχει ένα ρόλο και το ερώτημα πάει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το γνωρίζετε και τι κάνετε γι' αυτό. Και τι κάνει η Επιτροπή Μάλλον Εξωτερική Δράση για να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία. Ε, Παρομοίω. Για την αναθεώρηση δεν θα πρέπει να ξαναδούμε τι σχέσει που μα με του Παλαιστινίου, να μην υπάρξει μια τεχνική αναθεώρηση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ισραήλ, ώστε όλε αυτέ οι σχέσει να αποκλείουν τι επιχειρήσει και το οικονομικό όφελο τη περιοχέ του επικισμού. Και τελευταίο, μια από τι μεγαλύτερε νίκε για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα αυτά ήταν ε, το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του Δεκεμβρίου του 2016 το οποίο χρησιμοποίησε φρασιολογία που ήδη είχε χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το πρόθεσε αυτό, δεν το διαφήμισε. Να κάτι που θα μπορούσαν ε, να έχουν κάνει. Ανοίγουν δρόμοι για την ε, προαγωγή αυτών των διαφορετικών μέτρων διαφοροποίηση, όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα κάτι μέλη τη, αλλά και σε συνεργασία και με άλλα μέρη ε, τη όλη διαδικασία. Κάτι από την Αμερικανική Ήπειρο, από την Αφρική. Όλοι πρέπει να αναλάβουν εδώ τις ευθύνες τους και θα έλεγα για να ολοκληρώσω με κάποιες ε, τελευταίες παρατηρήσεις ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την ε, στάση και τη συμπεριφορά του business as usual σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Πρωθυπουργός Νοτανιάχου που θα έρθει εδώ τον ε, Δεκέμβριο νομίζω ότι περιμένει να λάβει χαιρετισμού και από τους 28 πρωθυπουργούς και αρχηγούς κατών κυβερνήσεων. Αλλά τι λέει αυτός προς, την, ε, προς όσους προειδοποιούν για την απομόνωση, για την τοποθέτηση του Ισραήλ διαφορετικά σε σχέση με τις διεθνείς του σχέσεις. Εν τέλει, για το Ισραήλ. Ο Ισραήλ είναι ο κατέχον και μόνο εκείνο μπορεί να αποφασίσει να πάυσει την κατοχή. Είναι μερικά πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κατημέλη για να ενισχύσουν τους Παλαιστινίους. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια διαδικασία συμφιλίωσης. Η Αίγυπτος έχει αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο, η ΙΠΑ φαίνεται να συγκατανεύουν έστω και από το παρασκήνιο, το αφήνουν και τα κράτη του κόλπου να εξελιχθεί και το Ιράν. Δεν λέω ότι αυτή η ειρηνευτική διαδικασία θα οδηγήσει σε αποτελέσματα, και μια κρίσιμη λύση μεταξύ ΦΑΤΑΡ και Χαμάς, αλλά αφήνει ανοίγματα για να γίνουν πράγματα να βοηθηθεί η λωρίδα της Γάζας. Απλά πράγματα. Την ε, ηλεκτροδότηση. Την άρση κάποιων από τους περιορισμούς για την πρόσβαση στη Γάζα. Πράγματα τα οποία έχουν επιδενωθεί από τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Γάζα. Θα ήταν και αυτός ένας τρόπος. Και να τελειώσω λέγοντας ότι το απαγορευτικό είναι οι διαχωρισμοί μεταξύ των κατομελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα ότι ενώ βλέπουμε να μην υπάρχει λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Βρυξελών, κάποια κάτι μέλη να συγκεντρώνονται σε ομάδες για να βρουν ε, αποτελεσματικούς τρόπους να υλοποιήσουν την δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν ε, εφαρμόζεται. Ε, είτε προς τη διαφοροποίηση είτε προς άλλα. Ίσως έτσι μπορέσει η ΕΚΠΑΤΗ πρόσωπος να εκπληρώσει την εντολή της. Και για να ολοκληρώσω, θα πρέπει και το Ευρωκοινοβούλιο να συνεχίσει να με τις ερωτήσεις του την κυρία Μογκερίνη για την ε, επίθεση ετικετών λόγου χάρη. Δεν μπορεί το Ευρωκοινοβούλιο να λάβει αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής αλλά μπορεί να έχει καταλητική δράση, το, τη δράση ενός καταλήτη στην γενικότερη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Για να σας πω κάτι ενθαρρυντικό, πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι ήταν. Από ό,τι ξέρω, Δεν μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση για τη Γάζα. Λόγω του, των φιλελεύθερων. Ε, ζητώ συγγνώμη απέναντι στα μέλη του, των φιλελευθέρων. Α, ο Ήβο, α πούμε, είναι φιλελεύθερο, φεύγει τώρα. Γιατί οι φιλελεύθεροι μπλοκάρουν αυτή τη συζήτηση. Είναι άθλια η κατάσταση. Το Ισραήλ είναι πανταχού παρόν εδώ. Είναι, κάνει λόμπι. Ακριβώ γι' αυτό η Παλαιστίνη είναι απούσα στι συζητήσει μα. Είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Είναι δύσκολο να κινητοποιήσουμε έστω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω να βελτιωθεί η κατάσταση. Πρέπει να βελτιωθεί. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους, να κάνω εγώ μερικές ερωτήσεις. Έχουμε διαβάσει πολλά συμπεράσματα του Συμβουλίου. Από το Συμβούλιο εξωτερικών υποθέσεων. Ε, αρκετά καλά. Αλλά γιατί δεν έχει δοθεί συνέχεια. Κάθε φορά που υπάρχει κάποια δράση, βλέπετε τώρα, ε, η Κύπρος, η Μάλτα, συγγνώμη, ε, κύριε Σιλικιώτη, αλλά φεύγουν σιγά σιγά. Η Ελλάδα, τι μπορούν να επιτύχουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, γιατί υπάρχουν. Και εδώ και 10 χρόνια είμαι μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κάθε φορά βγάζει συμπεράσματα το Συμβούλιο. Αλλά τι κάνουμε με αυτά τα συμπεράσματα, τι τα κάνουμε τα συμπεράσματα. Επίση, κατά την άποψή σα, ποιο είναι το όραμα του Ισραήλ για το όραμα. Γιατί ακόμα και τη λύση του ενός κράτους την φοβούνται. Ε, Ενό κράτου βέβαια που δεν θα, είναι, δεν θα προωθεί το apartheid έτσι, και που όλοι οι πολίτες θα έχουν τα ίδια δικαιώματα. Όταν συναντήσαμε τους ε, Ισραηλινούς ε, πολιτικούς και διπλωμάτες, δεν μα δίνουν ποτέ απαντήσει σε αυτό το θέμα του ενός ή δύο κράτη, α πούμε. Είναι γενική και αόριστη. Και δεν θέλω να πω ότι είναι καταθλιπτικό αυτό, αλλά φοβάμαι ότι συνεχίζουμε να έχουμε συμφωνίες, έχουμε τη συμφωνία για την αεροπορία. Δηλαδή, βασικά πληρώνουμε τους Ισραηλινούς για την κατοχή και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Και δίνουμε και λίγα λεφτά στους Παλαιστίνιους, έτσι, για να υπάρξει και κάποιος μετριασμός, ας πούμε, των επιπτώσεων της κατοχής. Ε, τα λεφτά μας είναι λεφτά μετριασμού των επιπτώσεων τη κατοχή. Λυπάμαι, είναι καταθλιπτικά όλα αυτά, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και τίμοι. Πρέπει να μιλήσουμε για το γεγονός ότι οι νέοι, ας πούμε, ε, είναι απόντες εκεί πέρα στην Παλαιστίνη. Ε, όσοι έχουν κάποια προσόντα λοιπά, φεύγουν. Δεν υπάρχουν, δεν μένουν στην Παλαιστίνη. Πρέπει επίσης να αναγνωρίσει η Ευρώπη ότι η κατάσταση αυτή είναι επικίνδυνη όχι μόνο για τους Παλαιστίνιους και τους ε, Ισραηλινούς, είναι επικίνδυνη για τους νέους ε, Παλαιστίνιους, ε, είναι επικίνδυνο και για τα κράτη-μέλη, γιατί βλέπουμε όλο και πιο εξαγριωμένους και απογοητευμένους ανθρώπους, ας πούμε. Βλέπετε, ας πούμε, ακόμα και στη Δανία, στη Δανία ε, καταλαβαίνουν οι δικοί μας νέοι, ας πούμε, ε, οι οποίοι μερικές φορές έχουν και ίδιοι προβλήματα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει να είσαι νέος, ας πούμε, στην Παλαιστίνη και να μην έχεις κανένα μέλλον. Ε, σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, συνεισφορές, οι οποίες ναι, με ήταν καταθλιπτικές, αλλά ήταν πάρα πολύ σωστές. Όσοι συνάδελφοι τώρα έχουν ερωτήσεις, παρακαλώ. Τους δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Ουκέν. Να υποφεληθώ από, την, από το γεγονός ότι έχουμε διακεκριμένους ομιλητές. Μιλούμε για μια παράνομη κατοχή και μιλάμε για διάφορους ε, παίκτες, για το Ισραήλ, για τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ξεχάσαμε κάποιον σημαντικό, που είναι η Σαουδική Αραβία. Δεν είπαμε κουβέντα για τη Σαουδική Αραβία. Έπαιξε ένα ρόλο μέχρι στιγμή, το ξέρουμε όλοι, αλλά ο νέος ε, πρίγκιπας, ε, από ό,τι ξέρω, προωθεί τη συμμαχία με το Ισραήλ. Την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του Γενικού Επιτηλίου Στρατού του Ισραήλ έδωσε μία ε, συνέντευξη σε μία ε, εφημερίδα ε, της Σαουδικής Αραβίας. Μην ξεχνάτε επίσης ε, το μπλοκάρισμα που υπάρχει στο Κατάρ γιατί δεν τους πήγε καλά αυτή η ιστορία. το πρόβλημα που υπάρχει με την Τουρκία και το μίσος Έχουμε την αίσθηση ότι η Ευρώπη, η Σαουδική Αραβία, το Ισραήλ και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μία ε, νέα συμμαχία για να σχεδιάσουν μια νέα μέση Ανατολή στα δικά τους μέτρα και σταθμά, με βάση τις δικέ τους επιθυμίες. Ε, από τη μία λοιπόν εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουμε λεφτά με το ένα χέρι ας πούμε και από την άλλη συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Κύριος μαχτά. Δεν θέλω να κάνω ακριβώς ερώτηση, αλλά μάλλον μια παρατήρηση. Οι τρεις ομιλητές, ο τελευταίος ειδικά ομιλητής, ε, ε, θα έχει πρόβλημα με αυτά που θα σας πω. Ε, για απλά λέω αυτά, έτσι. Ε, θα σας πούνε ότι είσαστε αντισημίτης με αυτά που λέτε. Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά πόσο υποκριτική είναι η ευρωπαϊκή πολιτική. Το είπατε με το δικό σας τρόπο, ευγενικά μερικές, φορέ, φορές, ότι λείπει ας πούμε η πολιτική βούληση κτλ. Αλλά υπάρχει πολιτική ε, υποκρισία από τα κράτη-μέλη. Είναι κατάφορη. Εξίσου υποκριτικό είναι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι, είμαστε απίστευτοι υποκριτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητώ συγγνώμη που είμαι τόσο όμω, αλλά παρότι δεν έχουμε την εξουσία που έχει το Συμβούλιο, για πολλά θέματα είμαστε συνομοθέτε. Οι συμφωνίε σύνδεση. Θα μπορούσαμε, τη συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ θα μπορούσαμε να την μπλοκάρουμε. Εσεί μίλησατε για το θέμα τη ετικετοθεσία για τα προϊόντα από του επικισμού. Σε ποιον βαθμό θα μπορούσαμε εμεί να απαιτήσουμε από την Κομισιόν την καλή εφαρμογή τη συμφωνία. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν απάτες. Αλλά ούτω ή άλλω είναι παράνομη αυτή η ιστορία και όλοι το ξέρουν. Η Κομισιόν το ξέρει, το Συμβούλιο το ξέρει και εμεί οι Ευρωβουλευτέ το ξέρουμε. Μην νομίζετε λοιπόν ότι είναι πιο υποκριτέ η Κομισιόν και το Συμβούλιο από εμά και από τι πολιτικέ ομάδε και το δικό μου και η δική μου πολιτική ομάδα. Υποκρίτρια είναι κι αυτή. Γιατί έχουμε πραγματικά ένα όπλο εντό αγωγικών, διπλωματικό όπλο, έτσι, για να πετύχουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αντιμετωπίζει τα, φα, λάθη και την υποκρισία της. Τα είπες και εσύ, Μάγκρετ. Έχουμε ε, τις συμφωνίες για τον ορίζοντα 2020 και το Ισραήλ συμμετέχει. Θα μπορούσαμε να αρνηθούμε να ψηφίσουμε τον προπολογισμό, αλλά ποιος θα τολμούσε να το κάνει αυτό. Επομένως, ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί υποκριτές, έτσι. Ε, ζητώ συγγνώμη, Μαγκρέτ, είμαι τόσο φλή και εσύ, έτσι. Είμαστε κι εμείς υποκριτές για να αλλάξουμε πολιτική θα έπρεπε ίσως να αλλάξουν οι πολιτικοί, έτσι. Το είπε ο Παλαιστίνιος φίλος. Αλλά καλό θα ήταν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φύγουν οι παλιοί πολιτικοί και να έχουν νέοι, φρέσκοι. Είμαστε μια ισχυρή μειοψηφία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως υπάρχει και μια ισχυρή μειοψηφία κρατών μελών. που καταγγέλουμε όλα αυτά τα πράγματα. Ζητώ συγγνώμη αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά είμαστε μειοψηφία. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα με τη δημοκρατία. Υπάρχουν μειοψηφίε. Ναι, Κλή, έχει το λόγο. Είμαι πολύ σύντομο. Ε, ακούω του συναδέλφου, βεβαίω με του συναδέλφου θα συζητούμε ε, τακτικά αυτά τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι εκφράζουμε και στην ίδια στι συνεδρίε τη αντιπροσωπείας ε, τα παράπονα μας, ε, την κριτική μας, κυρίως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το περασμένο ε, Φεβρουάριο επισκεφθήκαμε αποστολή της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου ε, την Παλαιστίνη, είδαμε από κοντά το τι συμβαίνει με την κατοχή. Ε, εκ μέρου τη Επιτροπή έστειλα εγώ επιστολή στην κυρία Μονκερίνη και ζήτησα μια συνάντηση για να ενημερώσω για το τι είδαμε και να ακούσω και τι δικέ τη απόψει, η οποία αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ. Είναι πολύ άσχολη η πάτη ε, αντιπρόσωπο. Ε, είπαμε θα την καλέσουμε στην Επιτροπή. Ε, Όμω παρόλα τα αυτά ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν διαφωνώ ποσό με τον ΕΤΟΑ, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Το Ευρωκοινοβούλιο, οι εξουσίε του, παρόλο που έχει κάποιε εξουσίε, είναι περιορισμένε. Ε, όμως, εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουμε ακόμα πιο έντονα. Να θέτουμε τα ζητήματα. Να φέρω ένα παράδειγμα. Η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους είναι ε, ένας βασικός στόχος και πρέπει να πιέζουμε και στην κατεύθυνση των κρατών και στην κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς ως Κοινοβούλιο αυτό που μας αναλογούσε το κάναμε. Τι κάναμε δηλαδή, αλλάξαμε πρώτα-πρώτα ε, αυτό μπορούσαμε... τον τίτλο τη ε, αντιπροσωπεία. Ναι, ναι. Η αντιπροσωπεία μα ήταν αντιπροσωπεία με το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Και έγινε αντιπροσωπεία με την Παλαιστίνη, όπω είναι όλε οι αντιπροσωπείε, για να καταδείξουμε ότι η Παλαιστίνη είναι κράτο. Και εγώ αυτό που ήθελα να πω στου. Ε, επειδή γίνεται αναφορά ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό που ήθελα να, να ζητήσω είναι ε, τι είναι εκείνο που μπορεί να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη Εμεί λέμε τακτικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο κύριο χρηματοδότη τη Παλαιστινιακή Αρχή και ταυτόχρονα ο μεγαλύτερο εταίρο. Ε, και έχει δίκιο ο Έντουαρ Μαρτίν όταν είπε ε, για τη συμφωνία σύνδεση. Ε, Βεβαίω, Έντουαρ, εγώ πολλέ φορέ στην Ολομέλεια η θέση τη ομάδα μου είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να απαγοποιηθεί η συμφωνία σύνδεση σαν ένα μέτρο πίεση. Αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω, αν υπάρχουν μέτρα συγκεκριμένα πίεση ε, τι λένε για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει εμπάρκο. Ε, είναι ένα θέμα που συζητιέται πολύ στο Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι όπω έγινε ε, για να αντιμετωπιστεί το άπαρχα τη Νοτιού Αφρική. Αυτά. Τελευταίος ομιλητής. Επίσης, εάν οποιοδήποτε από του προηγούμενου ομιλητέ, του προηγούμενου πάνελ θέλει να αυτές ερωτήσει, να τι ακούσουμε. Για να είμαι πολύ σύντομος, να συστηθώ, είμαι ο Μικέλ Βιέγκας. Είμαι μέλος του ΠΣΠ, του Πορτογαλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, από τα κόμματα που στηρίζουν τους Παλαιστινίους και τον αγώνα τους. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Ε, προβλέπετε να ξεκινήσει κάποια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της Συμφωνία Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ εφόσον κάποια νομολογία υπάρχει το Δεκέμβριο του 2016 το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κήρυξε παράνομη την ε, εφαρμογή τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκή Ένωση Μαρόκου λόγω της περιοχή της Δυτική Σαχάρα. Με αυτή την ομολογία υπόψη, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει μια διαδικασία παρόμοια κατά τρόπον ώστε να κηρυχθεί παράνομη οποιαδήποτε συμφωνία που θα αφορούσε τα παλαιστινιακά εδάφη που παρανόμως κατέχονται από το Ισραήλ. Ε, to We're talking here about... Εδώ μιλάμε ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Μιλάμε για κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία και συνένεση, δεν υπάρχει και τέτοια πολιτική. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν άλλου που έχουν εξωτερική πολιτική. Δείτε τι γίνεται στη Συρία. Οι Ευρωπαίοι ακολουθούν τη Ρωσία, το Ιράν, την Τουρκία. Ούτε καν τι είπα, Διότι είπα που απουσιάζουν επίση. Είναι θέμα ηγεσία εδώ, ηγετικού ρόλου και λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι όπως φαίνεται, δεν έχουμε μια εξωτερική πολιτική, έχουμε μια κοινή. Ε, χρειάζεται μια προσωπικότητα που να μπορεί να το κάνει αυτό πραγματικότητα. Να πείσει τα κάτι μελη Έχει συμβεί στο παρελθόν. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Το δεύτερο είναι ότι αν δείτε την ιστορία της Ευρώπης, και τη στάση τη παρέμβασή στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση. Αυτό που μπορούσε να γίνει με 9-10 χώρες, τώρα πια δεν γίνεται με 28. Κάποιες από τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίω από τι νέε. έχουν άλλη άποψη για το Ισραήλ ανάλογα με την ιστορία τους και τις ιστορικές τους σχέσεις. και τις εκφράζει περισσότερο τη του είναι ελεύθερη δημοκρατία του Ισραήλ παρά κάτι άλλο. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που μπορούμε να το έχουμε υπόψη. Το Κοινοβούλιο βεβαίω και πρέπει να ζητήσει από την είπατε εκπρόσωπο που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει και να καταθέσει τα όσα γνωρίζει επί του θέματος. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε σε αυτό, κάτι δεν λειτουργεί καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι τυπικότητα, θεωρώ. Το άλλο που είναι πολύ σημαντικό σε ό,τι αφορά το διεθνές δίκαιο και τη συμμόρφωση με τα ψηφίματα ασφαλείας του Συμβουλίου του ΙΕ είναι ότι δύο μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, τρία μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν πολύ στενές σχέσεις με το Ισραήλ. Ε, η η Ρωσία και η Κίνα. Η Κίνα επενδύει μαζικά στο Ισραήλ. Πολύ χρήμα ρέει προς τα εκεί. Οπότε θέλει να έχει συμβόλαια και συμβάσει η Κίνα εκεί. Ο δρόμος του μεταξιού. Καθόλου δεν την νοιάζει δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους και η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Κάποιος ανέφερε την προσάρτηση της Κρυμαίας. Ε, ναι. Είναι επίσης ένα παράδειγμα για το πας μια χώρα θεωρεί σωστό ότι μπορεί να μπει και να βάλει πόδι. Η απόφαση των Ευρωπαίων κάποιοι ανέφεραν την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα η σχέσεις ε, προς την Συρία και την Κύπρο, ιδίως σε, σχέση, σε θέματα ενέργειας κλπ, βαθαίνουν για τη Σαουδική Αραβία τώρα. Η Σαουδική Αραβία ζητά μια νέα εξισορρόπηση των δυνάμεων στην περιοχή. Αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ. Ο νέος πρίγκιπας ήδη απειλεί, απειλεί να αποσταθεροποιήσει την ίδια τη Σαουδική Αραβία. το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία έχουν κοινά στρατηγικά συμφέροντα, κοινέ ε, πληροφορίε στι μυστικέ του υπηρεσίε. Ήταν προφανέ εδώ και χρόνια. Και από τη Βαγδάτη οι μυστικέ υπηρεσίε πήγαιναν στο Ισραήλ για να ανταλλάξουν στοιχεία στο παρελθόν. Για τη Συρία, για το Ιράκ, για την Ιεμένη. Είναι μια πραγματικότητα που θα μείνει μαζί μα για πολύ καιρό. Πρέπει οι Ευρωπαίοι να ξυπνήσουν και να γνωρίζουν τι συμβαίνει. Γι' αυτό επέμεινα ότι δεν αρκεί να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ζητήματα αυτά, αλλά τα ίδια τα συμφέροντα που εκφράζουν οι Ευρωπαίοι σε αυτή την περιοχή και εκεί πρέπει να τα επεξεργαστούν διαφορετικά. Μόχλευση έχουμε, δυνατότητα άσκηση πίεση έχουμε. Πολλέ φορέ μίλησα στου υπευθύνου για το μόχλευση που διαθέτουμε. Το Ισραήλ δεν σέβεται το διεθνέ δίκαιο, όμω ε, έχουμε φτάσει εμεί να μην σεβόμαστε του δικού μα νόμου σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ μα συμφωνίε. Ναι, πρέπει λιγάκι να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου. Μπα τη ξυπνήσει κανεί, αλλά πρέπει οι Ευρωπαίοι, θεσμοί, κράτη, μεμονωμένα άτομα, όσοι συμμετέχουν σε think tank, να αναλάβουν δράση. Θα απαντήσω στα γαλλικά γιατί γαλλικά με ρωτήσατε. Η πρόεδρος έκανε μια πολύ σωστή παρατήρηση. Η κατάσταση στο Ευρωκοινοβούλιο δεν είναι αυτή που ήταν πριν από 10 χρόνια. Είναι μια παρατήρηση που μας θλίβει, μας στενοχωρεί. Τα ελπίζαμε να συνέβαινε το αντίθετο. Το Ευρωκοινοβούλιο να καταλάβαινε περισσότερο, να αντιλαμβανόταν περισσότερο την οξύτητα του προβλήματος και το κίνδυνο για την ειρήνη στη Μεσόγειο και την όλη περιοχή. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαβε να είναι ενεργός, να έχει συνείδηση της αρνητικής εξέλιξης των πολιτικών πραγμάτων και για τα ερχόμενα χρόνια. Αυτό που διαπιστώνω προσωπικώς, κατοικώντας εδώ και 50 χρόνια στο Βέλγιο, είναι ότι τη δεκαετία του 60, 80% των Βέλγων ήταν υπέρ του Ισραήλ με την Ιντιφάδα του 87 άνοιξαν τα μάτια τους, όχι μόνο των Βέλγων αλλά των Ευρωπαίων και ανακάλυψαν τη φροκαλαιότητα της κατοχής και την, ε, ε, τον εξευτελισμό που επιβλήθηκε στον Παλαιστινιακό λαό. Αυτή η συνειδητοποίηση μετά το 87 επέτρεψε στους ευρωπαϊκούς ε, θεσμούς να στραφούν λίγο πιο σοβαρά προς το Παλαιστινιακό ζήτημα και Το 1985 προσεκλήθη η Παλαιστινιακή Αρχή να ε, συμμετάσχει σε όλα τα μεσογειακά ε, προγράμματα, όπως τη διαδικασία της Βαρκελόνης, την πολιτική γειτονία του 2004, την πολιτική για την, ε, για την Βόρεια Αφρική. Εκλήθη η Παλαιστινιακή Αρχή και το Ευρωκοινοβούλιο συνέταξε μια σειρά από εκθέσεις με πολύ καλές συστάσεις ήταν η δεκαετία του 90, αρχές του 2000. Το 2005 λοιπόν έχουμε πάλι την εντύπωση ότι υπάρχει υποστοχώρηση. Ή παναχώρηση μάλλον. Πρώτα απ' όλα εγώ ίδιος διαπιστώνω κόποση. Κόποση από μια σύγκρουση που διαρκεί εδώ και πολλά χρόνια. Και που δεν διαφαίνεται καμία πιθανή λύση. Δεύτερον, από την διεύρυνση του 2004 είναι προφανές. Δέκα νέες χώρες οι διαφωνίε και οι διαχωρισμοί στην Ευρώπη έχουν πλέον έρθει στο φω. Οι χώρε τη Ανατολική Ευρώπη, όπω την Παλαιστίνη, έχουν μια στάση πολύ ε, λιγότερο ξεκάθαρη από κάποιε χώρε τη Δυτική Ευρώπη. Τρίτον, υπάρχει ένα πολύ ισχυρό λόμπι υπέρ των Ισραηλινών που δρά εντό του Κοινοβουλίου, που δρά εντό των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, εντό τη κοινωνία των πολιτών. Το είδαμε και σήμερα κιόλα και η Ευρώπη έχει πει ξεκάθαρα δεν θα τιμωρήσουμε το Ισραήλ. Δεν υπάρχουν κυρώσεις για το κράτος του Ισραήλ γιατί είναι μεγάλος εμπορικός εταίρος. Και είναι επίσημη δήλωση αυτή. Η Ευρώπη που σήμερα έχει τη δυνατότητα να ασκήσει κάποιο είδους επιρροή για το Ισραήλ δεν την ασκεί. Για τον πολύ απλό λόγο ότι εντός των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων δεν υπάρχει σύγκληση απόψεων. Το βλέπουμε, το είδαμε στην πληροφορία της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ το 18. 14 χώρε ψήφισαν υπέρ της Παλαιστίνης, 13 κατά, κάποιες απήχαν και υπήρχαν ε, και αποχές. Το είδαμε και στην UNESCO. Το έχουμε δει επανειλημμένος. Όλα αυτά έχουν κάνει να υπάρχει τώρα πιστοχώρηση της αλληλεγγύης. Όχι στο επίπεδο του κόσμου των πολιτών, σε επίπεδο θεσμών. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη απόκληση μεταξύ των θεσμών που υποτίθεται ότι εκφράζουν του ευρωπαϊκούς λαού και των ίδιων των πολιτών που είναι οι ευρωπαϊκοί λαοί και έχουν πολύ πιο προοδευτικέ, πολύ πιο προηγμένε θέσει για την πραγματιστική κατανόηση τη όλη κατάσταση. Και τώρα ο λόγο στον κύριο Λόβατ. Μας τελειώνει και ο χρόνος. Όταν ήθελες να θέσεις και εσύ ερωτήσεις, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να σου δώσουμε το λόγο. Έχουμε μόνο 10 λεπτά. 5. Γιατί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων έχουν πέσει σε φωνές βόντος εν γιατί συνειδητοποιούμε ότι αν ξανανοίξουμε θέματα τα οποία έχουμε κλείσει, μπορεί να μην τα ξανασυμφωνήσουμε. Επομένω, οι θέσεις οι οποίες τα μέλη, ακόμα και αυτά που συμφώνησαν το 2012, μπορεί αν τα ξανασυζητούσαμε τώρα, να μην συμφωνούσαν τα μέλη, δηλαδή τα κράτη-μέλη. Και στην πραγματικότητα αυτό θα εξέθετε την διαίρεση των κρατών μελών, αφενός. Από την άλλη, Υπάρχει μια νομική και πολιτική εντολή από το 2012 και με ψηφίσματα και τα λοιπά για να κάνουμε διάφορα πράγματα. Καταρχάς, να, να εφαρμοστεί σωστά η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τα προϊόντα από τους επικισμούς. Υπάρχει μια νομική και πολιτική εντολή για την Κομισιόν και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να κάνουν κάτι, χωρίς να χρειάζεται να επανέλθουμε για να... στο Συμβούλιο δηλαδή για νέα συμπεράσματα. Το θέμα είναι πώς θα υποστηρίξουμε και θα πιέσουμε και θα σπρώξουμε την ύπατη εκπρόσωπο να κάνει κάτι και να αισθάνεται ότι έχει την υποστήριξη και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ένα, ενός μεγάλου αριθμού κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά το Ισραηλινό όραμα, ε, το εργατικό κόμμα μέχρι στιγμής είναι αυτό το οποίο έχει πιο λεπτομερή ε, σχέδια για το που πάει η χώρα. Και δεν είναι ένα όραμα για δύο κράτη μέχρι ε, στιγμής. Είναι μονομερής ε, διαχωρισμός ή μονομερή ειρήνη, το λένε πολλά πράγματα. Αν το κοιτάξετε όμως το πλάνο του εργατικού κόμματο, είναι μια επισημοποίηση της σημερινή πραγματικότητα. Δηλαδή ουσιαστικά ξαναμετακινούμε τα έπιπλα του Τιτανικού που έλεγα πριν. Και το να ριζώσει η ιδέα του ενός κράτους τελικά. να κρατήσει το στρατιωτικό έλεγχο στα εδάφη που κατέχει, τα Παλαιστινιακά δηλαδή. Υπάρχει μια κριτική από την ε, δεξιά του Ισραήλ, ότι η δεξιή πολιτική δεν ήταν τόσο έτσι καλή στο να περάσουν το νέο όραμα για το Ισραήλ όσο ήταν η πολιτική του εργατικού κόμματος. η ε, πολιτική που προωθεί η δεξιά σήμερα είναι η πολιτική που ξέρετε, ε, αυτή που βλέπετε. Ε, δεν θέλουν να αλλάξουν τίποτα. Θέλουν να προωθήσουν την ίδια κατάσταση, να τη διαιωνίσουν κτλ. Και το είπε και ο Νετανιάχου. Έχει γράψει και ένα βιβλίο. Δεν υπάρχει τίποτα μυστικό σε αυτά που σα λέω. Ποια δυσκολία έχει ο Νετανιάχου. Δεν έχει καμία δικαιολογία να τον κρατάει πίσω με τον Ομπάμα και την προηγούμενη Αμερικανική κυβέρνηση ε, μπορούσε να πει «Α, αν είχαμε ένα καλύτερο Αμερικανό πρόεδρο θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, ας πούμε, με, με τους επικισμούς κτλ». Τώρα έχει έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος και αυτό κινείται προ τη δική του κατεύθυνση. Το θέμα είναι λοιπόν γιατί δεν πάει ακόμα πιο μακριά ο Νιτανιάχου. Υπάρχει πολλή πίεση ε, από, την, ε, από τα δεξιά του κόμματό του να πάει ακόμα πιο μακριά και γίνεται λόγο στην νομοθεσία ε, όλο και περισσότερο για επέκταση των ε, επικισμών. και για ρύθμιση της ε, περιουσίας των Παλαιστινίων. Σιγά σιγά κινούνται λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιος είναι ο ρόλος των Σαουδαράβων. Το όραμα των Σαουδαράβων. Ποιος είναι ο ρόλος των Σαουδαράβων. Τι χρειάζεται η Σαουδική Αραβία. Είναι να τονώσει το στρατόπεδο που είναι κατά του Ιράν. Στην πραγματικότητα συντάσσεται με το Ισραήλ, ας πούμε, για να ενισχύσει τη δική του, ασφα... τη δική του ασφάλεια. Τουλάχιστον εγώ έτσι ερμηνεύω τα γεγονότα. Ο πρίγκιπας θεωρεί ότι είναι ένας ε, μοντέρνος ηγέτης και θέλει να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ. Στην πραγματικότητα δεν πάει τόσο μακριά όσο πήγαινε ο προκάτοχός του. Ε, τώρα, για να τελειώσω, για τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, Συμφωνία Σύνδεσης, δεν είμαι εμπειρογνώμονας, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί πάρα πολύ σκέψη, ούτως ώστε να Υποβάλλουμε σωστά το ερώτημα στο δικαστήριο. Γιατί αν θέσουμε λάθος το ερώτημα στο δικαστήριο, δηλαδή με μια λάθος διατύπωση πούμε, του αιτήματο, μπορεί να πάμε πίσω χρόνια. Το δικαστήριο, μην ξεχνάτε, με τις αποφάσεις του παίζει σημαντικό ρόλο ε, για να αποκλειστούν τα προϊόντα από τους επικισμούς ε, στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Με τι αποφάσει του δικαστηρίου αποφάσεις παλιές, πριν από 10 χρόνια και παραπάνω. Ε, στην πραγματικότητα είχαν ζητήσει η εξαγωγή στο Ισραήλ ε, προσέφηκαν στο δικαστήριο για να ε, δικαιωθούν και να μπορούν τα προϊόντα τους να παραμείνουν ε, στη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να θέσουμε στο δικαστήριο σωστά την ερώτηση. Μια λάθος διατύπωση θα μας πάει πίσω. Πολύ ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πολύ σημαντικές, όραμα και έμπνευση παρεμβάσεις σας. Απαριθμίσαμε όλα τα εμπόδια. Παρόλα αυτά, παρότι εστιάσαμε πολύ στα εμπόδια, διαφέρονται κάποιες προοπτικές. Αυτό που είναι αλήθεια είναι ότι και οι δύο λαοί έχουν αλλάξει. Υπάρχει μια μετάβαση στην οτροπία των ανθρώπων ε, και όχι μόνο στην περιοχή, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε διάφορες χώρες, στην Τσεχία και σε άλλες χώρες, ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν μία δίκαιη λύση. Γιατί δεν κάνουμε περισσότερα. Ε, δεν θα το έλεγα έλλειψη δημοκρατίας. Εν πάση περιπτώσει, έχω... Θέλω, θα ήθελα να σταματήσω τίποτα εδώ με αυτή τη νότα και να σας ευχαριστήσω όλους. Ήταν μια πολύ σημαντική διάσκεψη. Παρότι, παρότι βγάλαμε τα πλητά μας στη φόρα. Πρώτος ευχαριστή και τους διερμηνείς.